Καλό σας απόγευμα. Θα ήθελα να αρχίσουμε με τις εργασίες μας. It's open. There is the red light. Yeah. Ah, okay. Allora, abbiamo al punto prima l'ordine del θα ήθελα καταρχήν να εγκρίνουμε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τους συναδέλφους, θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Περνάμε στην εξέταση ορισμένων σημείων της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να πληροφορήσω τους συναδέλφους και ζητώ συγνώμη διότι εξαιτία τεχνικών ε, προβλημάτων στο σύστημα διανομής κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, στην αρχή αυτής της εβδομάδας δεν ε, διαβιβάστηκαν όλοι οι φάκελοι στους συναδέλφους. Ελπίζω να επιληθεί αυτό το θέμα σήμερα. Διαφορετικά, ε, όπως σας είπα, δεν εξαρτάται από εμάς. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την ψηφοφορία σε σχέση με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε 60 τροπολογίες, τις οποίες και θα ψηφίσουμε. Στη συνέχεια έχουμε εντάξει το φάκελο για την Equitable Life, την ασφαλιστική. Ζητήθηκε από τους συναδέλφους Βίλαντ μακίνες να ενταχθεί αυτό το θέμα, γιατί η αναφορά έχει παραμείνει ανοιχτή, εκρεμής. Άρα θα πρέπει εμείς να γνωμοδοτήσουμε επί του σημείου αυτού. Μετά θα ακούσουμε του συναδέλφου Βόλης και Χέφνερ για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών και θα μας μιλήσουν για την έκβαση της συνάντησης που είχαν με τους συνεισηγητές της ΑΦΚΟ. Θα ήθελα να σας πω εκ των προτέρων ότι η Επιτροπή ΑΦΚΟ θα συναντηθεί στις 13 Δεκεμβρίου το βράδυ στο Στρασβούργο για να ορίσει, να επικυρώσει την συμφωνία. Ε, Επίσης έχουμε τα σημεία 8, 11, 13 και 14. Ως προς τις αναφορές ε, για την ελευθεροτυπία στη Ρουμανία θα ήθελα να σας πω ότι πέρα από τους ετούντες θα είναι παρόντες και ορισμένοι Ρουμάνοι από τις αρχές ο κύριος Μανιού που είναι υπεύθυνο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ε, Τούρκαν και Γκαλέα που είναι νομικός σύμβουλος. Αυτό αφορά το σημείο 18. Το σημείο 2 αφορά την έγκριση των πρακτικών της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου και της 25ης στις 6 Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τους συναδέλφους, θεωρώ ότι εγκρίνονται τα δύο αυτά πρακτικά. Εγκρίνονται νομίζω. Σας υπενθυμίζω ότι προσαρτάτε στην ημερήσια διάταξη και τα σημεία Β, το τμήμα Β, όπου εγγράφονται οι αναφορές οι οποίες θα πρέπει να κλείσουν. Εάν δεν υπάρξει μια διαφορετική παρέμβαση από κάποιο συνάδελφο, θα εγκριθούν και θα αρχιοθετηθούν κατά αυτόν τον τρόπο, στο τμήμα Β, μέσα στην προθεσμία των εργασιών της Επιτροπής μας. Δεν έχω άλλες ανακοινώσεις, αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, Περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης και αρχίζουμε με την ψηφοφορία σε σχέση με τη γνωμοδότηση για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπα... του... της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συμβουλίου και Επιτροπής. Ah, με συγχωρείτε. Χάνκης. Νομίζω ότι είχαμε πολλές ε, ευκαιρίες να αλλάξουμε τις ε, απόψεις μας, γι' αυτό προτείνω να αρχίσουμε με τις εργασίες μας, εφόσον δεν επετεύχθη κάτι τέτοιο. Αρχίσουμε με την ψηφοφορία λοιπόν. 14, τοπολογία 14. Θα έχουμε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση, ερωτάτε, Όχι, διανατάσεως και θα γίνει έλεγχος μόνο αν χρειαστεί. Μπορούμε να κάνουμε έναν ε, δοκιμαστικό έλεγχο αν το επιθυμείτε. Sì, prego. Πρόεδρε, δεν έχω κάρτα μαζί μου για να ψηφίσω. Ας γίνει μία δοκιμή. Uh, Και να γίνει καταμέτρηση. Βεβαίως ε, θα γίνει καταμέτρηση, αλλά ας κάνουμε μία ε, δοκιμή για το ηλεκτρονικό σύστημα. Αρχίζουμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία στο άρθρο 2 υπαριθμών 14 τη συναδέλφου Όκιν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 15 στο άρθρο 2. Υπέρ παρακαλώ. Καταπίπτει, γιατί εγκρίθηκε η προηγούμενη τροπολογία, η 14. Γιατί δεν εγκρίθηκε, με συγχωρείτε, λέει η Πρόεδρος. Καταπίπτει, διότι απορρίφθηκε η τροπολογία 14. Έκανα εγώ λάθο, λέει η πρόεδρο. Τροπολογία 1 στην παράγραφο 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 στο άρθρο 3 στοιχείο α υπέρ. Κατά. Αποχές Θα χρειαστεί να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. So Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 στο... Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 στο άρθρο 3β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 στο άρθρο 4 παράγραφος 1 α υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 στο άρθρο 4 1 δέλτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 στο άρθρο 4, παράγραφος 2, γάμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 στο άρθρο 4, υπέρ, α, καταπίπτει. 6 all'articolo 4. 6 υπέρ στο άρθρο 4 σημείο δέλτα κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο ε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 άρθρο 4 παράγραφος 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 21 στο άρθρο 4 παράγραφος 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 σε ξεχωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Δεκτή. Ξέχασα τις αποχές, λέει η πρόεδρος. Δεκτή η τροπολογία. Τροπολογία τώρα επτά Καταπίπτει 23 άρθρο 4 παράγραφος 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 24 στο άρθρο 5 παράγραφος 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25 στο άρθρο 5 παράγραφος 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 στο άρθρο 5 παράγραφος 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 στο άρθρο 5 παράγραφος 3 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 στο άρθρο 7 παράγραφος 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τις υπόλοιπες να τις δούμε όλες μαζί. Συλλογικά. Δέκα Όλες οι υπόλοιπες τροπολογίες σαν με ενιαία ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Άρα ψηφίσουμε Ηλεκτρονικά τελική ψηφοφορία. Ε, Εγκρίνεται με 17 ψήφους με τον συνάδελφο που δεν έχει κάρτα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Χάνκης. 17, σας ευχαριστώ συνάδελφοι για την εργασία σας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κάσμαν γιατί ήταν πολύ διαλλακτικός και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Χάνκης. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι το 6 Δίνω το λόγο στον Ετούντα. Στον κύριο Braithwaite. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνετε για να ενημερώσω την Επιτροπή Αναφορών ε, για αυτήν την ε, μακροχρόνια περιπέτεια. Είμαι ο Πολ Μπάιτμιτ και έρχομαι από την IMAC. Ε, πρόκειται για μια ομάδα δράση των μελών τη Equitable Life, 40.000 μέλη που πληρώνουν εισφορέ. Shame the disgraceful of the British Treasury. Ε, τα θύματα της Equitable Life είναι ένα εκατομμύριο και ε, πάνω από 12.000 ε, Γερμανοί και Ιρλανδοί πολίτες. Πρώτη φορά ε, η αναφορά υπευλήθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από έξι χρόνια και το έκανα αυτό γιατί ε, το Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών ε, δεν ε, μπορούσε να εξετάσει απαρκώς το ζήτημα της κακής διαχείρισης Equitable Life. Πρέπει να πω ότι η αδιάλακτη στάση έχει συνεχιστεί η και μάλιστα και με την ε, νέα κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν ε, δύο κόμματα. Από ό,τι γνωρίζω υπήρξε μια ειδική επιτροπή Equitable Life στην ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έγιναν συγκεκριμένες παρουσιάσεις και η Diana Wallis παρουσίασε μια έκθεση 350 σελίδων η οποία εγκρίθηκε ε, με συντριπτική πλειοψηφία. Η βασική σύσταση ήταν να κληθεί η Βρετανική κυβέρνηση και ε, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δεχθούν και να εφαρμόσουν ε, σωστά όλες τις συστάσεις ε, του, του ε, κοινοβουλευτικού διαμισολαβητή του Ηνωμένου Βασιλείου. Όμως η Μεγάλη Βρετανία αγνόησε παντελώς τη συγκεκριμένη έκθεση. Επίσης αγνόησε οποιαδήποτε προσπάθεια από ευρωβουλευτές, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως επίσης και από τον προηγούμενο πρόεδρο της Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που εκδόθηκε η έκθεση του Βρετανού διαμισολαβητή στο Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει της οποίας ε, οι Βρετανοί ρυθμιστές και ε, το Υπουργείο Οικονομικών ήταν υπεύθυνοι τεράστιας ρυθμιστικής ανεπάρκειας ε, και επίσης αποφασίστηκε ότι, ενώ είχε αποφασιστεί ότι έπρεπε να αποζημιωθούν τα θύματα απορρίφθηκαν μάλιστα τα πορίσματα του, του, του διαμεσολαβητή και στη συνέχεια ένας ε, δικαστής που δεν είχε πια ε, καθήκοντα διορίστηκε για να γίνει κάποια αποζημίωση μόνο προς τα μέλη που ε, είχαν υποστεί τεράστιες ζημίες. 18 μήνες πήρε η όλη διαδικασία και η έκθεση έγινε μετά από τις πρόσφατες εκλογές του Μαΐου. Όμω, βασικά στοιχεία έχουν παραμείνει ίδια και συνεπώς δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η αποζημίωση που, που προτείνεται είναι μόνο 400.000 ευρώ διαδικασία στο τέλος εγκαταλείφθηκε ε, με, χωρίς να ανταποκριθεί στο ύψος των περιστάσεων. Στις 20 Οκτωβρίου ε, ήταν η χειρότερη, 20, 20 Οκτωβρίου ήταν η χειρότερη ημερομηνία για μας που προσπαθήσαμε να αποζημιωθούμε γιατί ήταν τμήμα της περιεκτικής ε, ε, έκθεσης για την μείωση των δαπανών. Ήταν πραγματικά μια μέρα πάρα πολύ κακών μαντάτων για μας. 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ ε, αποζημιώσεων έπρεπε να καταβληθούν σε μια τριετή περίοδο με επιπλέον 6 εκατομμύρια ευρώ ε, σε πολλές, ε, επί πολλές ε, δεκαετίες θα έπρεπε να πληρωθούν σε συνταξιούχους. Αυτό είχε συσταθεί η Βρετανική κυβέρνηση είχε δεχθεί να ακολουθήσει τη μεθοδολογία του δικαστή ότι ήταν 5,2 εκατομμύρια οι ζημιές, όμως η ΙΜΑΚ εκτιμά ότι είναι περίπου 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ τελικά οι ζημιές. Τώρα, τα παραποιημένα ε, έγγραφα του Υπουργείου ε, ισχυρίζονται ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν είναι πολύ λιγότερες ε, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΆΙΜΑΚ μόνο το 1 τέταρτο των αποζημιώσεων θα καταβληθούν τελικά. Ε, δεν υπάρχει δεν, ε, η, η κατανομή ε, των αποζημιώσεων ε, δεν είναι καθόλου λογική. 37.000 συνταξιούχοι, ένα πέμπτο, κατά το ένα πέμπτο θα αποζημιωθούν. Τι καταπληκτική λύση. 10.000 ε, πιο ηλικιωμένοι συνταξιούχοι που βρίσκονται στην ηλικία των 80 τώρα και που ξεκίνησαν την σύνταξή τους, ε, τις φορές τους πριν από το 1992 δεν θα λάβουν απολύτω τίποτα ω αποζημίωση και αυτοί είναι οι άνθρωποι που είναι οι πιο ευάλωτοι και οι πιο ηλικιωμένοι. Ένα εκατομμύριο θύματα θα μοιραστούν 930 εκατομμύρια ε, σε μία περίοδο τριών ετών. Αυτό είναι 15% των πραγματικών ζημιών που υπέστησαν. Αυτή δεν είναι η δικαιοσύνη για την οποία αγωνιστήκαμε τόσο πολύ ούτε στο περιεχόμενό τη, ούτε και στην ε, κατανομή των αποζημιώσεων. Η κυβέρνηση δικαιολογείται λέγοντα ότι είναι πάρα πολύ κακή η κατάσταση τη Βρετανική οικονομία και θεωρεί ότι το ζήτημα έχει καλυφθεί ε, ικανοποιητικά και ότι πρέπει να ε, το ξεχάσουμε. Όμως έγινε μια υπόσχεση από την κυβέρνηση συνασπισμού για δίκαιη και διαφανή ε, αποζημίωση προς ε, τους κατόχους ε, ασφαλιστηρίων και μάλιστα πολλοί βουλευτές είχαν οι ίδιοι υποσχεθεί στις περιφέρειές τους να υποστηρίξουν και να ε, υπερψηφίσουν τη σωστή αποζημίωση των θυμάτων του σκανδάλου της Equitable Life. Ελπίζω να μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο αισθάνονται προδομένα τα μέλη της ΣΥΜΑΚ ε, από την κυβέρνηση αυτή, όπως και από την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί αυτό που προτείνεται ε, είναι εντελώς παράλογο και ε, πενιχρό δεν ε, έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα εκείνων που με δυσανάλογο τρόπο υπέστησαν ε, ζημιές. Η ΕΜΑΚ ξεκίνησε μία αναθεώρηση σε βρετανικό κα δικαστήρια και η επιχειρηματολογία της είναι ότι γίνεται κακός υπολογισμός ε, κατά 45% ε, της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί και ότι αυτό είναι ενάντια στην υπόσχεση της Βρετανικής κυβέρνησης ότι 10.000 ε, συνταξιούχοι παρέμειναν χωρίς απολύτως καμία αποζημίωση. Είναι πραγματικά θλιβερό ότι πρέπει και πάλι να ε, πάμε στα δικαστήρια την καινούρια μας κυβέρνηση όταν ε, η διαδικασία του διαμεσολαβητή σκοπό έχει να αποδίδει δικαιοσύνη με, με διαφανή τρόπο. Και οι επενδυτές, οι Γερμανοί και οι Ιρλανδοί που δεν γνωρίζουν τίποτα και που παραγνωρίζονται συνεχώ, ε, είναι γεγονός ότι επειδή δεν είναι Βρετανοί υπήκοοι, δεν θα πρέπει να ε, διέπεται το καθεστώς του από το 85% της αποζημίωσης γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή είναι προσωρινά, έχει πτωχεύσει η Βρετανική κυβέρνηση. Έπρεπε όμως να έχουν δικαίωμα να μπορούν να βασιστούν στους Βρετανούς ρυθμιστές. Θα έπρεπε να ε, λάβουν 100% αποζημίωση και όχι μόνο 85%. Η ΜΑΚ έχει συμπεριλάβει στο σκεπτικό της ε, ενώπιον του δικαστηρίου ότι κάτι τέτοιο πρέπει να ισχύσει και για τους μη Βρετανούς υπηκόους. Όμως ο κύριος Όσμπορν ανακοίνωσε στις 20 Οκτωβρίου ότι θα βοηθήσουμε και εκείνους που βρίσκονται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και που έχασαν χρήματα λόγω της κατάρρευσης της Equitable Life. Θα ήθελα να ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα να να διαφωνήσει με το προφίδιο Σάλμπιμ to την πονηρά αλβιώνα ε, και να μπορέσει να αγωνιστεί υπέρ την αποζημίωση των συνταξιούχων ε, και ενάντια στην κακοδιαχείριση των Βρετανών ρυθμιστών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή, στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Η Επιτροπή τρέφει κάθε κατανόηση για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι Βρετανοί πολίτε που έχουν χάσει τα εισοδήματά του λόγω τη κρίση του Equitable Life. Θα θέλαμε ωστόσο να υπογραμμίσουμε ότι οι οδηγίες για την ασφάλιση ζωής και τομέων εκτός τη ασφάλισης ζωή οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιβάλλουν ε, αποτελεσματικά συστήματα διευθέτησης διαφορών εξοδικαστικός στα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια παλιά ιστορία. Και η μόνη δυνατότητα που θα είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή θα ήταν να εκκινήσει τη διαδικασία επί παραβάση. Καθώς όμως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παγίως αποφασίζει με την ομολογία του, η επιπαραβάση διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αποκατάσταση υφισταμένου, ε, αποκατάσταση της ευθυγράμμισης υφισταμένου, επαναλαμβάνω, υφισταμένου ε, εθνικού δικαίου με το ευρωπαϊκό όχι όμως για να αποκατασταθούν ζημιές από προηγούμενη ασυμβατότητα του εθνικού με το ευρωπαϊκό δίκαιο που εντωμεταξύ έχει αντιμετωπιστεί. Η Επιτροπή θα ήθελε να σας διαβεβαιώσει ότι, αν, ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση αυτή και αν προκύψει αδίποτε ένδειξη παραβίασης, παράβασης του ευρωπαϊκού δικαίου είναι διεθμένη να αναλάβει δράση και να παρέμβει. Αυτά είναι τα σχόλια που μπορούμε να σας προσφέρουμε πλευρά της Επιτροπής προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον Πολ Μπρέτουιθ για την ε, παρουσία του εδώ και για την ε, τοποθέτησή του απέναντι στι Επιτροπές των Αφορών. Ω πρώην πρόεδρος της Επιτροπής, της Επιτροπής, Ερευνητικής Επιτροπής ε, για το Equitable Life, λυπούμε που χρειάστηκε να ξανάρθετε εδώ. Ήλπιζα ότι θα έχει ολοκληρωθεί και προ ικανοποίηση των ετοιμάτων σας το ε, θλιβερό αυτό το θέμα, θλιβερή αυτή η υπόθεση. Δυστυχώ όμω ακόμη δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα. Ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι από την Επιτροπή που όμω έχει δει το Equitable Life εδώ και πολλά χρόνια, ίσω να μην είναι ενήμεροι για τι λεπτομέρειε τη υπόθεση αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τι είδου δράση θα μπορούσαμε να λάβουμε από πλευρά τη κοινοβουλευτική μα Επιτροπή. Εμένα αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερω είναι ότι πολλοί από του συναδέλφου έχουν λάβει ε, ατομικά κάποια επικοινωνία από τα θύματα που βλέπουν ότι δεν είναι ικανοποιημένα από τη ρύθμιση που έχει δοθεί στο σε επίπεδο ε, Ηνωμένου Βασιλείου, οι μέτοχοι, οι, αυτού του εξωτικού συστήματος. Και για δε την ετοιμιγορία του δικαστή Osborne της 28 Οκτωβρίου, επαναλαμβάνω το κείμενο, που λέει ότι θα πρέπει όσοι από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν χάσει χρήματα λόγω της ε, πτώχευσης Equitable Life να ε, στηριχθούν νομίζω ότι το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το θέμα αυτό, διότι υπάρχουν δικαιούχοι μάλλον εξωτικών ταμείων και μέτοχοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουν πληγεί. Και πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί κάθε πρόσφορη αποζημίωση για όλα τα θύματα ανεξαρτήτως της υπηκότητάς τους. Δεν ξέρω όμω αν αυτό έχει επιτευχθεί. Έχω αποστείλει βεβαίω ω μέλο του Κοινοβουλίου, αλλά προσωπικά στο όνομά μου δηλαδή ε, τη σχετική επιστολή ε, στο Υπουργείο των Οικονομικών, αλλά δεν έχω λάβει καμία απάντηση και έτσι δεν είμαι σε θέση να σα ενημερώσω. Πάντω χαίρομαι ότι η που η ευκαιρία που μα δίνεται επιτρέπει να συζητηθεί τουλάχιστον το θέμα εδώ σήμερα. Όταν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, στόχο μα ήταν να στηρίξουμε τα θύματα και όσους αποδεικνύονταν πως είχαν πέσει θύματα στην ε, εξέλιξη αυτής της διαδικασίας. Και επίσης βλέπαμε ότι ήταν και πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες μας και η δυνατότητα να βοηθήσουμε σε κάποια αποκατάσταση των ζημιών. Εάν υπάρχει λοιπόν τη δυνατότητα, πρέπει να μεριμνούμε τουλάχιστον εμείς όσοι έχουν την ευθύνη για την αποκατάσταση των σημειών να το πράττουν κατά τρόπο ικανοποιητικό και προς όλα τα θέματα. Φαίνεται όμως δυστυχώς ότι ακόμη αυτό δεν έχει εξασφαλιστεί. Και πάλι λοιπόν, όσο και να με θλίβει το ότι είστε εδώ για αυτό τον λόγο σήμερα, ευχαριστώ που ήρθατε και ελπίζω μέσα από τη συζήτηση να, έχουμε, να καταλήξουμε σε ένα πρόγραμμα δράσης, σε κάποιες αποφάσεις ε, μετά τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ η κυρία Γόλης έχει το Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και κυρία Μαγκίνες, και εγώ βέβαια έχω εμπλακεί πολύ στην υπόθεση αυτή. Με μεγάλη μου θλίψη βλέπω τον κύριο Μπρέιθουιτ και πάλι εδώ, αν και πάντα με χαρά τον βλέπω, αλλά όχι για τέτοιους λόγους και από αυτές τις συνθήκες. Γιατί και εγώ όπως και πολλοί άλλοι ελπίζω ότι θα μπορούσαμε να επιλύσουμε το θέμα αυτό μέσα από τις, νέες, από τις της ε, ε, κυβέρνηση συνασπισμού, που θεωρούσαμε ότι θα είναι πιο δεκτική στα αιτήματά μας. Φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια πρόοδος, ε, δηλαδή η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως ε, τα πορίσματα στα οποία έχει καταλήξει ο διαμεσολαβητής, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει και στην σχετική δράση για την αποκατάσταση των ζημιών. Εγώ προσωπικώς ζήτησα διαβεβαιώσεις τουλάχιστον για τα θύματα που δεν διαμένουν στο Ρήμανο Βασίλειο και έλαβα ανεπίσημα τη διαβεβαίωση ότι θα αντιμετωπιστούν και οι δικές τους περιπτώσεις. Θα ήθελα όμως να έχω μια πιο ε, επίσημη, πιο δημόσια δηλαδή διαβεβαίωση στη διάθεσή μου και ελπίζω να μπορέσει να ε, πιέσει προς αυτήν την κατεύθυνση η Επιτροπή μας. Επίσης, για τον κύριο Braithwaite, ε, θα ήθελα να επισημάνω ότι πολύ σωστά επισημαίνει πως είναι άνισο το σύστημα με το οποίο προσφέρεται αποζημίωση. Αυτό έχει επισημάνει εξ αρχής και το έχουμε δει και εμείς τα τελευταία χρόνια όπου διαπιστώνεται αφενός μεν στο Ηνωμένο Βασίλειο να καταραίουν φερρυπίν οι Ισλανδικές τράπεζες όπου αμέσως αποζημιώθηκαν οι παθόντες ενώ στην Equitable Life τους είχαν αφήσει ε, μετέωρους ε, επί σειρά ετών. Και τώρα βλέπουμε ότι ακόμη δεν έχει δοθεί η κατάλληλη και έγκαιρη αποζημίωση. Ανησυχώ λοιπόν, αλλά δεν αρκεί να ανησυχούμε. Πρέπει να βρούμε μια πρακτική μέθοδο που θα σήμαινε, πιστεύω, έτοιμα προς τη νέα κυβέρνηση για μια σαφή δημόσια δήλωση ή ενδεχομένω να προσκαλέσουμε κάποιον από την νέα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για να απαντήσει στις ερωτήσεις καταρχάς για τις ευρωπαϊκές πτυχές, δηλαδή το πώς καλύπτονται οι ε, παθόντες που δεν ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεύτερον και πώς θα δοθεί μια ισότιμη αποζημίωση, μια δίκαιη αποζημίωση στους ε, παθόντες του Ηνωμένου Βασιλείου. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2011 θα αρχίσουν να αποζημιώνονται κάποιοι. κάποιοι. Ευχαριστώ, πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Πολ Μπρέιθουιτ και τον συγχαίρω κιόλα ε, γιατί εξακολουθεί να ασκεί πίεση. Ε, από την αρχή το έκανε, πριν από 7 χρόνια, όταν για πρώτη φορά ήρθε να μας δει και τότε εγώ ήμουν πρώτος αντιπρόεδρος της ε, ε, επιτροπής αυτής και είχα προτείνει ειδική επιτροπή για να εξετάσει το θέμα η οποία πραγματικά ε, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά και αμερόληπτα υπό την ηγεσία της κυρίας Μακίνες. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά στο Δουβλίνο συγκεκριμένα ε, άνθρωποι που είχαν επενδύσει καλή πίστη και θεωρούσαν ότι προστατεύονταν από τον νόμο απογοητεύτηκαν τελικά ε, τους πρόδωσε ο νόμος, δεν υπήρχε καμία προστασία. Ε, και έπρεπε να ε, συνεχίσουν οι δικαστικέ διαδικασίε. Είναι μια πάρα πολύ κακή κατάσταση, απαράδεκτη. Κανένα πολιτικό κόμμα δεν, ε, ε, δεν αντέδρασε αξιοπρεπώς στην όλη διαδικασία και πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει αυτό το θέμα. Εγώ ψήφισα μαζί με άλλου, υπέρ όλων των συστάσεων, ανεξαρτήτως με το μπορούσαμε να τι καταπιούμε ή όχι, να είναι αποδεκτέ από όλα ε, τα ενδιαφερόμενα μέρη και ε, του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και των ε, αναφερόντων και κανένας τελικά δεν τήρησε τις υποσχέσεις του και μιλάω και για την κυβέρνηση των εργατικών την προηγούμενη του Ηνωμένου Βασιλείου. Εντάξει υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες και πάντοτε μπορούν να γίνονται πολιτικές δηλώσεις σχέση με αυτό αλλά πραγματικά Μιλάμε για τεράστια ποσά, είναι ε, κάτω από 3 εκατομμύρια λίρες και πριν από μερικές ημέρες ε, 6 ε, δισεκατομμύρια ε, ε, ήταν μια συμφωνία του Ηνωμένου ε, Βασιλείου ε, με την Vodafone και δεν μπορούμε να δώσουμε 3 εκατομμύρια λίρες για να αποζημιώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και υπάρχει βέβαια και η εμπειρία της Ισλανδίας. Βέβαια ότι και οι άνθρωποι αυτοί δεν έπρεπε να είχαν αποζημιωθεί γιατί τότε είχαμε να κάνουμε με οικονομική κατάρρευση και η αδράνεια θα είχε προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή. Δεν θέλω δηλαδή να συγκρίνω τη μία κατάσταση με την άλλη γιατί δεν είναι διαφορετική δεν, δεν είναι η ίδια κατάσταση. Καταλήξαμε σε διεξοδικά συμπεράσματα στο πλαίσιο τη Ειδική Επιτροπή. Οι συστάσει έγιναν αποδεκτέ, εγκρίθηκαν και νομίζω ότι αν έρθουμε σε επαφή με τη Βρετανική κυβέρνηση, που όπω γνωρίζει ο Ρότζερ ε, δεν ε, ε, λατρεύει ιδιαίτερα τα, τους, ε, το κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου ούτε τα διάφορα όργανα που υπάρχουν τα ρυθμιστικά. Ε, κάτι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να αποζημιώσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους ε, στους οποίους υποσχέθηκαν αποζημίωση γιατί διαφορετικά μία ακόμη φορά θα ε, μιλάμε για μια κυβέρνηση που έχει εξουσία χωρίς, καθόλου, χωρίς να έχει καθόλου αρχές και εγώ παραμένω ε, στη διάθεση της ΆΙΜΑΚ και του ε, Paul ε, για την ε, δικαστική αναθεώρηση και πιστεύω ότι ως κοινοβούλιο πρέπει να ε, δούμε τι θα γίνει και με τους Ιρλανδούς και Γερμανούς ε, αναφέροντες, ε, οι οποίοι και εκείνοι πρέπει να λάβουν αποζημίωση και δικαιοσύνη σε σχέση με τις αξιώσεις τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να συμφωνήσω και εγώ εν γέννη με τους συναδέλφους που μίλησαν νωρίτερα, δεν θα τα επαναλάβω. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πράγματα τα οποία έχουμε δει ήδη στις εκθέσεις, ε, στην έκθεση της Ειδικής Επιτροπής. Είδαμε ότι δεν δόθηκαν οι αποζημιώσεις όπως έπρεπε, δεν αντιμετωπίστηκε δηλαδή το πρόβλημα όπως έπρεπε. Εγώ θα ήλπιζα η διαμεσολαβήτρια του Ηνωμένου Βασιλείου να έχει έρθει σήμερα εδώ για να μας εξηγήσει περισσότερο αυτή την υπόθεση. Με ενθαρρύνει βέβαια για να αισιοδοξία το γεγονό ότι είναι κάποιο πιο θετικά διακείμενη στην υπόθεση αυτή η νέα ε, βρετανική κυβέρνηση. Αλλά καλό θα ήταν να δούμε για τη διαμεσολαβήτρια τη Βρετανίδα να μα δώσει πιο συγκεκριμένε πληροφορίε. Γι' αυτό παρακαλώ το θέμα αυτό να το διατηρήσουμε στην ημερήσια διάταξη και να το ξανασυζητήσουμε όταν θα έχει και, την, ε, και, και η διαμεσολαβήτρια την ευκαιρία να έρθει εδώ στι Βρυξέλλε για να συζητήσουμε μαζί τη αυτά τα πράγματα. Να μην το κλείσουμε δηλαδή σήμερα το θέμα ε, Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να παρέμβει. Δεν ξέρω κατά πόσο ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, θέλει να απαντήσει. Ο κύριος Μπραιτ ε, θα ήθελα σεβόμενος στην Επιτροπή να πω το εξής. Ε, αν είχαμε ακολουθήσει την, την ε, υπόδειξη της Επιτροπής 7 χρόνια πριν, δεν θα χρειαζόταν να συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή. Βεβαίως μας δεσμεύουν οι συνθήκες και το κοινοτικό ακτιμένο, αλλά όταν πρόκειται για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών υπήρχε μία δεοντολογική αρχή. Τώρα υπάρχει μία νομική αρχή και είναι η χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η συνθήκη της Λισαβόνας. Αναγνωρίζω αυτά που είπε η Επιτροπή. Δεν με εκπλήσει, αλλά η Επιτροπή έδρασε ανεξάρτητα από τη γνώμη του Επιτρόπου 7,5 χρόνια πριν. Θέλει ο να προσθέσει κάτι άλλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαρία Μαγκίνες, την Νταϊάννα Βόλις και τον Μάικλ Κάσμαν ε, για τα καλά τους λόγια. Ε, ένα αριθμητικό στοιχείο λάθος έκανε. Τρία δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια λίρες. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μπερδέψει κανείς ε, την τάξη των αριθμών. Αλλά είναι γεγονός ότι είναι εύκολο να λέει κανείς ε, πω, πόσο καιρό έχει καθυστερήσει όλη η διαδικασία, πρέπει να παραμείνει στην ημερήσια διάταξη Επιτροπής των Αναφορών. Ε, κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει αποζημίωση, αυτό είναι το βασικό. Γι' αυτό φτάσαμε στην διαμεσολαβήτρια για ε, αποζημίωση. Ελπίζω, Σερ Άμπραχαμ, να ακολουθήσει τις συστάσεις σας ε, και να επισκεφθούν και εκείνοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να παρίσταμε και εγώ όταν ε, κάτι τέτοιο προγραμματιστεί την επόμενη χρονιά. Σε σχέση με αυτό που είπες, Νταϊάννα, οι καταβολές θα αρχίσουν να γίνουν ε, το καλοκαίρι του 2011 για μια περίοδο τριών ετών, αλλά δυστυχώς όχι νωρίτερα. Θα ήθελα παρόλα αυτά να ευχαριστήσω τους Ευρωβουλευτές και το Προεδρείο της Επιτροπής που ε, με προσκάλεσαν. Ε, ε, Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να σταματήσουμε εδώ. Αυτή είναι η άποψη, η ομόφωνη άποψη της Επιτροπής. Απλώς θα πρέπει να δούμε ποια είναι και τα όρια της δυνατότητας παρέμβασής μας. Θα πρέπει να στείλουμε τις γνωμοδοτήσεις και τις συστάσεις για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αποστείλουμε όλα αυτά τα στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας και όπως είπε ο κύριος Κάσμαν να μην αποσταλεί σε κάθε βουλευτή χωριστά αλλά στον πρόεδρο του σώματος έτσι ώστε να ε, γνωρίζουν αυτά τα δεδομένα όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου και να μιλήσουμε και στον πρόεδρό μας, τον κύριο Μπούζεκ, ο οποίος θα μπορούσε να αποστείλει μια επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων. Αυτά είναι τα δεδομένα και Εάν συμφωνείτε, κλείνουμε με αυτή τη συζήτηση, αλλά αφήνουμε ανοιχτό. Α, η συνάδελφος Μαγκίνες ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι, εγώ συμφωνώ με τις προτάσεις σας. Υπάρχουν τρία τμήματα. Το πρώτο είναι οι συστάσεις, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι. Όμως υπάρχουν δύο ακόμη ζητήματα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά ε, τους ε, μη Βρετανούς κατόχους ασφαλιστηρίων συμφωλέων. Χρειαζόμαστε περισσότερη δράση για το θέμα αυτό και άμεσα μάλιστα. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακούσαμε διάφορα ότι όλα καλά θα πάνε, αλλά αν δεν είναι αυτό γραμμένο κάπου, τότε ε, λέμε στους ε, ε, στις περιφέρειές μας κάτι το οποίο δεν ξέρουμε αν ισχύει. Χρειαζόμαστε κάτι γραμμένο, κάτι σε χαρτί. Δεν ξέρω, θα έρθουν στη, στη, στην επόμενη συνεδρίασή μας να μας απαντήσουν σε ορισμένα ερωτήματα ε, κατά, πόσο το πακέτο της αποζημίωσης αφορά όλο τον κόσμο. Και επίσης υπάρχει και το πρόβλημα της ανισότητας μεταξύ των διαφόρων κατόχων των, ε, των ασφαλίσεων. Αλλά πρέπει να το θεωρήσουμε ένα ευρωπαϊκό θέμα, γιατί αυτό θα βοηθήσει πολύ την ε, στην ε, ε, δουλειά της. Νομίζω ότι πρέπει να εστιαστούμε πολύ περισσότερο σε αυτό το ζήτημα από εδώ και στο εξή. Νομίζω ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι ως προς αυτό το θέμα θα πρέπει να ζητήσουμε μια πρωτοβουλία από τις εθνικές αρχές, δηλαδή στα, στην ανακοίνωσή μας θα εντάσσεται και αυτή η ιδέα, δηλαδή να δούμε ε, πώς ο καθένας μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του. Εντάξει. Άρα θα αποστείλουμε ακριβώς όπως προτείναμε αυτά τα δελτία. Ευχαριστώ τον Ετούντα και περνάμε στο σημείο 7 που είναι η πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο είτε στον κύριο Χέπνερ είτε στην κυρία Wallace. Η κυρία Γουόλης. Okay, ναι. okay, then uh, ξεκινήσω εγώ, θα μιλήσω γερμανικά, αν μου επιτρέπετε. Ναι, και έχουμε εδώ τους γερμανείς μας. Τις τελευταίες εβδομάδες η δουλειά για την έκθεσή μας ε, και εμβαθύνθηκε και επιταχύνθηκε με την πολύ επιτυχημένη συνεργασία που είχαμε και με τους κοιόδης ηγητές μπορέσαμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις. Τη Δευτέρα η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων συζήτησε και την Τρίτη έλαβε την απόφασή της για την έκθεσή της. Εχθές δε το απόγευμα εμείς μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου προσπαθήσαμε σε πανατριμερή διάλογο να επιλύσουμε τα ακόμη εκρεμή ζητήματα. Μας διευκόλυνε σε αυτή την ε, συνομιλία το γεγονός ότι τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε πάντοτε παγίως υπογραμμίσει το περιθώριο χειρισμών και είχαμε διερευνήσει το περιθώριο χειρισμών και των άλλων πλευρών. Το Συμβούλιο βεβαίως εμένει στην ε, δική του μεθοδολογία λήψης αποφάσεων και τα κράτη-μέλη με δυσκολία δέχονται ε, τροποποίησεις σε ορισμένα σημεία για τα οποία ενημερωθήκαμε και για τα οποία είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη μπορούν να αλλάξουν στάση. Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά επιτυχημένοι σε αυτό το τριμερή διάλογο. Το αποτέλεσμα μας φέρνει αρκετά κοντά στην πρόταση της Επιτροπής. Δηλαδή, πρώτον, ο αριθμός των κρατών μελών από το 1 τρίτο, τα 9 δηλαδή, ε, έχει μειωθεί στο 1 τέταρτο, δηλαδή 7 κράτη-μέλη, αυτά τα οποία αντιτίθενται στην πρόταση αυτή. Μεγάλη επιτυχία του Κοινοβουλίου. Επίσης, η παράλογη και άσχετη με την πραγματικότητα ε, επαλήθευσης με βάση 300.000 υπογραφές ε, θα ξεκινήσει από την Επιτροπή εφόσον η πρωτοβουλία ξεκινάει από, 5, ε, από 7 διαφορετικές πλευράς, από 7 διαφορετικά κράτη-μέλη. Αυτά είναι άλλη μια μεγάλη επιτυχία μα που ζητούσαμε εδώ και καιρό. Αυτό το οποίο δεν καταφέραμε και που ζητούσε η Επιτροπή των Αναφορών ήταν να επιβάλλουμε τη δυνατότητα να υποβάλουν τέτοιου ε, να υπογράφουν τέτοιου είδους ε, πρωτοβουλίες όχι μόνο πολίτες, δηλαδή ηθαγενείς των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και αλλοδαπή που διαμένουν νόμιμα, αυτό το καταφέραμε, και επίσης δεν καταφέραμε και να μειώσουμε την ηλικία για την συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία ε, της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας στα 16 χρόνια που θέλαμε ισχύει το έτος της νομιμοποίησης όπως γνωρίζετε στα, ε, που ισχύει στα κράτη-μέλη για την εξφράση του δικαιώματος του εκλέγην. Ένα άλλο ζήτημα ήταν αυτό των προσωπικών δεδομένων. Ξέρετε ότι για να υπογράψει κανείς μια ε, τέτοια πρωτοβουλία πολιτών θα πρέπει να δίνει και στοιχεία διαβατηρίου, αριθμό διαβατηρίου ή αριθμό, αριθμό ταυτότητα. Όμως εμείς λέμε ότι αυτό πράγμα δεν μπορεί να είναι νόμο και σύμφωνο με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δεδομένου δε ότι σε ορισμένε χώρες δεν υπάρχει το σύστημα της ταυτότητας, ε, δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό αυτό. Εδώ λοιπόν το Συμβούλιο συζήτησε εντατικά αυτήν την υπόθεση. Κάποια κράτη που ζητούσαν εξάπαντος τον αριθμό ταυτότητας ε, υποχώρησαν, παρέμειναν όμως κάποια τα οποία είπαν ότι πρόκειται για όρο εκτρώνου κάνευ και θέλουν οπωσδήποτε ορισμένα λίγα κράτη ένα ε, με την καταγραφή του αριθμού ταυτότητας του υπογράφοντος. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε στη λύση να υπάρχει υποχρεωτικά σε όλη την Ευρώπη το όνομα η διεύθυνση, η υπηκότητα, η ημερομηνία γεννήσεως και η υπογραφή ως απαιτούμενα για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή σταθερά για να μπορούν όλα τα κράτη-μέλη να επαληθεύσουν. Και αυτό που δεν έγινε δεκτό ήταν να συμπεριλαμβάνεται και ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας ή, το, τα στοιχεία των, ε, τα ονόματα των ε, ε ανιόντων ε, πατέρας, πατέρα και μητέρας δηλαδή. Αυτά δεν θα καταγράφονται. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα Α η οποία έχει δεχθεί αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα ως Ευρωπαϊκή Σταθερά, υπηκότητα, ημερομηνία γεννήσεως, όνομα, υπογραφή και τα άλλα κράτη που είναι πιο απαιτητικά έχουν ένα χωριστό ε, έντυπο στο οποίο μπορούν να ζητούν αριθμό ταυτότητας και τα λοιπά. Και συμφωνούμε στα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα για τον υπογράφοντα. Αυτά είναι τα ελάχιστα που απαιτούνται σε όλα τα κράτη-μέλη και δεν είναι υποχρεωμένο κανένα κράτος να, να ζητήσει επιπλέον στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο βρήκαμε μια λύση. Επίσης, δεν μπορέσαμε παρότι υπήρχε κάποιο άνοιγμα από πλευρά Συμβουλίου αλλά και Επιτροπής να προχωρήσουμε ως προς το 18 μήνο της διάρκειας. Και το άλλο, το σχετικό με την συλλογή των υπογραφών online. Ήταν ένα θέμα στο οποίο βρήκαμε αντιμετωπίσουμε πάρα πολλέ ε, δυσκολίες. Η οικονομική υποστήριξη αλλά και η διαφάνεια ιδιαίτερα έχουν ε, κατά βάση ε, λυθεί ως εξής. Ως προς την διαφάνεια θέλουμε να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα του ποιος υποστηρίζει μια ε, τέτοια πρωτοβουλία πιο τη χρηματοδοτεί και κάθε ε, εισφορά άνω των 500 ευρώ πρέπει αυτόματα να δημοσιοποιείται. Αυτό δηλαδή ε, το όριο το οποίο έχουμε και για τα έσοδα των ευρωπαϊκών κομμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τα άλλα, υποχρεούται να προσφέρει την αρρωγή της, δηλαδή να έχει ένα help desk, να το πω έτσι, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς το λένε όμως, δεν το λένε helpdesk αυτοί. Α, contact point, σημείο επικοινωνίας, έχει σημασία, ε, κατ' ουσία είναι το ίδιο πράγμα με ένα helpdesk, ε, για την θέση εφαρμογή αυτού του συστήματος. Ήταν ένα δύσκολο θέμα στις διαπραγματεύσεις. και προτιμήσαμε να υποχωρήσουμε ε, ώστε να κερδίσουμε κάποια άλλα σημεία ως ε, προς την ε, περίοδο της εισαγωγής του συστήματος. Υπήρχαν κάποια κάτι που μας είπαν ότι δεν θα μπορούσαν μέσα σε έξι μήνες να είναι έτοιμα, αλλά ούτε καν στους 12 και βέβαια δεν μπορούσαμε ούτως άλλως να επιβάλλουμε κυρώσεις σε κάποιο κράτος το οποίο θα ήταν έτοιμο εγκαίρος για να αν είχαμε επιβάλει το χρονικό διάστημα των έξι μηνών. Τουλάχιστον όχι μέσω αυτού του κανονισμού, αυτής της ρύθμισης υπήρχαν άλλα έμεσα μέσα κυρώσεων, αλλά πάντως όχι άμεσα. Τελευταία παρατήρηση, η ιδέα της δημόσιας ακρόασης, που ήταν ίσως και το κύριο σημείο, το κύριο διακύβευμα εδώ, ποιος θα ακούσει τι έχουν να πούν οι πολίτες, ποιος θα αξιολογήσει αυτό το ένα εκατομμύριο υπογραφές, πώς θα φτάσουν μέχρι το κοινοβούλιο ή αν θα έρθουν με τη μορφή μιας επιστολής κτλ. Λοιπόν, προσπαθήσαμε ε, η Επιτροπή θέλει να μην είναι υποχρεωτικέ οι ακροάσει, αλλά κατά περίπτωση να κρίνεται εάν πρόκειται να γίνει ακρόαση ή όχι. Εμεί αυτό που καταφέραμε ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ισότιμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να το πω έτσι, να αποφασίζει, να είναι αρμόδιο δηλαδή, για τη διεξαγωγή τέτοιων ακροάσεων. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε, εκμεταλλευόμενη το γεγονό ότι θα ανατίθετο αυτή η αρμοδιότητα για τη λήψη απόφαση για την ακρόαση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να απαλλαγεί τον δικό τη ευθυνών. Ε, αυτό το αντιμετωπίσαμε, το αποτρέψαμε και τελικά είμαστε ισότιμοι και στην υποχρέωση αλλά και στα δικαιώματα. Στην υπόθεση αυτή. Μπορεί να μην αναφέρεται λοιπόν ρητά η φράση μέσω της αρμοδίας επιτροπής, δηλαδή της Επιτροπής Αναφορών, ξεκάθαρα, ε, το κοινοβούλιο λαμβάνει και τα λοιπά την απόφαση, αλλά ε, όσο και αν δεν αναφέρεται ρητά μέσα στο κείμενο, είναι σαφές το ποια είναι η Επιτροπή αρμόδια, ποια είναι η Επιτροπή η οποία θα ε, δει την πρωτοβουλία αυτή των πολιτών, τις ένα εκατομμύριο υπογραφές που έχουν συλλεγεί και που θα αποτελέσει και την το φόρουμ στο οποίο θα γίνει η συζήτηση, η ακρόαση, όπως είπα, από κοινό μαζί με την Επιτροπή. Εν τέλει και συνολικά νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Ξέρω ότι κάποια προβλήματα δεν τα λύσαμε όπως τα θέλαμε. Ήταν κάπως επώδυνες διαπραγματεύσει. Ξέρω ότι και η Νταϊάννα σε ορισμένα σημεία δεν είναι ευχαριστημένη. Σε ορισμένα όμως μπορούμε να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Η συνάδελφος η κυρία Γουόλης θέλει το λόγο. Νομίζω ότι έχει δίκιο ο Γκέραντ. Είναι εκπληκτικό για μένα να κάθομαι εδώ και να ακούω τον κατάλογο και να τότε συνειδητοποιώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει πραγματικά βάλει ένα σήμα κατά τεθέν ε, στην σχετική νομοθεσία και νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι για τη συμμετοχή της ε, συγκεκριμένης Επιτροπής γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος ε, δεν είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με μερικά πράγματα αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές θα είναι πολύ καλύτερο μέσο σε σχέση με αυτό που είχαμε αρχικά ε, ως πρόταση, όπως επίσης ε, και σε σχέση με την πρώτη, τον καρπό της πρώτης επεξεργασίας ε, του Συμβουλίου. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο φιλικό προς το χρήστη, πολύ πιο χρήσιμο. Οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη διαδικασία. Δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος άλλος θα ήθελε το λόγο και πάλι ο συνάδελφος. Εάν δεν αν δεν γίνει συζήτηση, ήθελα να πω ότι είχαμε αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ε, και με τη συνάδελφο Νταϊάννα Γουόλες και με τους συνεισηγητές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά σας και για τη δυνατότητα να παρισφρήσετε και να μπορέσετε να συζητήσετε ε, τροπολογίες συμβασμού των γραμματέα, των David Law και τους άλλους συνεισηγητές της ΑΦΚΟ. Ήμασταν ε, πολύ ε, επιτυχής εξαιτία της σοβαρής συνεργασίας από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σας ευχαριστώ όλους. Χωρίς μικρόφωνο. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές γιατί ήταν εξαιρετική η εργασία με απτά αποτελέσματα και θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτή την κοινή προσπάθεια. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω την ετοιμότητα των μελών της Επιτροπής Αναφορών να συνεργαστούν για ένα προσχέδιο το οποίο ε, οδηγούσε σε πολλά ερωτηματικά. Και βλέπουμε σήμερα ότι σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα ήμασταν συνενετικοί. Αυτό είναι ενθαρρυντικό και εντυπωσιακό και έτσι εμείς οι βουλευτές μπορούμε να εργαστούμε όταν μας απασχολεί μια τόσο σοβαρή ευρωπαϊκή υπόθεση. Και πάλι να σας συγχαρώ για την εξαιρετική αυτή συνέργαση. Δεν νομίζω ότι κανείς άλλος θέλει να παρέμβει, φαίνεται πως όχι. Και εγώ ευχαριστώ με τη σειρά μου τους συναδέλφους Hefner Wallis για αυτή την ε, συνεργασία. Παρά τους ε, ιονούς καταφέραμε πολλά πράγματα ως προς το ρόλο της Επιτροπής μας και σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, διότι όταν ε, ξεκινήσαμε αυτή τη μάχη για τον ρόλο της Επιτροπής μας, πολλοί προσπάθησαν να αποψηλώσουν αυτές τις προσπάθειες, την προσπάθεια δηλαδή των εισηγητών, των σκιωδών και προσπάθησαν να αποτελέσουν ένα ανάχωμα για τις εργασίες μας. Όμως είχαμε ένα πολύ ε, στενό χρονοδιάγραμμα και εσείς τα καταφέρατε μέσα στα πλαίσια του περιορισμένου χρόνου. Χαίρομαι διότι δεν υπάρχει πια καμία σκιά ως προς την εργασία σας και την εργασία μας και απέστειλα ε, ένα υπόμνημα προς τον πρόεδρο Μπούζεκ για να αλλάξει ο κανονισμός και να μπορούμε να οργανώνουμε και ακροάσεις μέσα στα πλαίσια της θητείας μας. Έτσι θα φτάσουμε σε ένα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα και μια μεγάλη νίκη. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η αναφορά στο σημείο 8 του κυρίου Ντεμπόνης και θα του δώσω το λόγο αμέσως για να παρέμβει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι διότι ότι μπορείτε να με ακούσετε ως αναφέροντα των Ιταλών εκτροφέων όπου μιλάνε για το, για το δίκαιο που αφορά το αντιτράστε και το, το Σύνταγμα της Ιταλίας. Εκπροσωπούμε τους Ευρωπαίους πολίτες στην, ε, στα κοινοτικά όργανα και βλέπουμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε να μειώσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα. Γι' αυτό σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε ευκαιρία να σας μιλήσω για την αμηχανία και απογοήτευση των εκτροφέων μας είτε από πλευρά στάσης του, της ταλικής κυβέρνησης είτε από πλευρά στάσης αντιτράστ προσπαθήσαμε να αποτανθούμε και στη Γερουσία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα μας αυτό της εκτροφής κουνελιών. Έχουμε να κάνουμε με έναν τομέα όπου δεν έχουν εφαρμοστεί οι οδηγίες και οι κανονισμοί από το Υπουργείο μας. Αυτή η παρελκυστική τακτική παραβιάζει τα άρθρα 41 και 42 του συντάγματος μας και δεν μπορούμε να φτάσουμε και στους στόχους της Ένωσης όπως ορίζεται από το άρθρο 3 της Συνθήκης. Θα θέλαμε ο θεματοφύλακας να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτή την ε, κατάσταση η οποία οδηγεί σε μια μεγάλη απογοήτευση. Όμως δεν εισακουστήκαμε και θεωρούμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί τι το, να εφαρμοστούν τα άρθρα 101 και 102 της συνθήκης. Η Ένωσή μας αντέδρασε αυτόνομα και θα θέλαμε να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ε, προέβησε μία ανακοίνωση, γιατί έχουμε απογοητευτεί. Θεωρούμε ότι δεν μπόρεσαν τα κοινοτικά όργανα να εγγυηθούν την εφαρμογή των κανόνων αντιτράστ. Στην ε, Ιταλία υπάρχει μία πολιτισμική καθυστέρηση σε σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς και την συμμετοχή τους. Γι' αυτό και δεν μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στους κανόνες ανταγωνισμού υπό την ευρεία έννοια. Αντιμετωπίσαμε πολλά εμπόδια και αυτό επιδίνωσε την κατάσταση της Ένωσής μας. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης και στα θεσμικά όργανα και θα σας εξηγήσω γιατί. Το πρώτο καμπανάκι το ακούσαμε το 2002 μετά από μια κοινοποίηση της Εθνικής μας Ένωσης και μία βασική καταγγελία. Τότε ήδη έπρεπε να καταλάβουμε ότι η αγορά δεν λειτουργεί σωστά, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για στρεβλωτική λειτουργία των χρηματιστηρίων εμπορευμάτων. Το 2009 η Επιτροπή ερεύνησε αυτό το δίκτυο όπου δεν υπήρχε διαφάνεια και ε, πλήττεται και ο ανταγωνισμός. Στην ανακοίνωση αυτή έφτανε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εποπτεία των αγορών. Μετά από 7 χρόνια η Ένωσή μας έκανε μια πρώτη καταγγελία με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις που ήταν ε, όμως ανεπαρκής για να αρχίσει μία διαδικασία έρευνας. Και θεωρήσαμε ότι υπάρχει μία κατάσταση κατάχρηση στην αγορά. Δηλαδή, θεωρούμε ότι δεν μπορέσαμε να φτάσουμε σε μία προανακριτική φάση για να δούμε κατά πόσο θα πρέπει να γίνει μία επίσημη προσφυγή. Προβήκαμε λοιπόν σε μία έρευνα και είδαμε ότι υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία που όμως όταν αναφέραμε στην αρμόδια αρχή, αντί να τους πείσουμε, ε, είδαμε ότι προσπάθησαν να συρρυκνώσουν τα αιτήματά μας. Θα έπρεπε λοιπόν οι καταναλωτές να υπομισθούν το τελικό τίμημα θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να μην δεχτούμε τα συμπεράσματα του αντιτράστ. Γιατί σε στιγμές ε, κρίσης θα πρέπει να μην υπάρχει παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού. Διαφορετικά φτάνουμε σε ολιγοπόλια ή μονοπόλια. Η Επιτροπή μίλησε για τιμές αγοράς χωρίς να δει πώς λειτουργούν τα καρτέλ και τι επιπτώσεις υφίσταται ο καταναλωτής. Όμως και πάλι δεν άρχισε μια ερευνητική διαδικασία. Αυτό μας οδήγησε στο να αποτανθούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη συνέχεια στην Επιτροπή Αναφορών. Θα πρέπει λοιπόν να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί που έχουν μεγάλη επίπτωση στην εφαρμογή της ε, κοινοτικής ρύθμισης. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν οι αρχές αυτές ή δεν πρέπει να προσφύγουμε στις ε, εθνικές, στην εθνική ένωμη τάξη. Εάν δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει της ε, επικουρικότητας. Περιμένουμε λοιπόν την περιμένουμε λοιπόν την απάντηση των ε, Ιταλικών αρχών. Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι έχουμε να κάνουμε με μια κρίση την οποία θα έπρεπε να αποφύγουμε, διότι δεν τηρήθηκε το Σύνταγμα και δυστυχώς πολλοί εκτροφείς και σφαγεία έπρεπε να σταματήσουν την εργασία τους. Πολλοί είναι υπερχρεωμένοι και δυστυχώς οι τράπεζες έχουν κατασχέσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πολλοί δεν μπορούν να πληρώσουν τα γραμμάτια που έχουν αναλάβει και είναι υπερχρεωμένοι. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και, την, και τους βασικούς κανόνες αξιοπρέπειας που ε, ορίζονται από την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει κατάφορη παραβίαση του κοινοτικού δικαίου διότι έχουμε να κάνουμε με μορφές εμπορίας των ατομικών δικαιωμάτων και τελικά οι καταναλωτές πρέπει να καταβάλουν το αντίτιμο διότι πρόκειται για δημιουργία καρτέλ τα οποία δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς το ε, κοινό καλό το οποίο θα πρέπει να διέπει όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Διότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δώσουμε έναν αγώνα επιβίωσης. Αυτό αφορά και τους εκτροφείς και τους καταναλωτές. Δεν αμφισβητείται όμως η νομιμότητα ορισμένων ενώσεων που προσπαθούν να μονοπολίσουν τις αγορές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με λειτουργία συγκεκριμένων λόμπι. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτός, αυτούς τους κανόνες και να λάβουμε υπόψη τις ρυθμίσεις αντιτράστ έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε αυτόν τον ε, αυταρχισμό. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στις ΗΠΑ προωθείται αυτό το δίκαιο του πλέον φτωχού μέσα στα πλαίσια των κανόνων αντιτράστ. Βλέπουμε όμως ότι εδώ στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ε, κυρώσεις και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κολλήσει στον τοίχο την ε, Ιταλία, διότι το χρηματιστήριο εμπορευμάτων δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, δυνάμει των ρυθμίσεων αντιτράστ και δυστυχώς δεν υπερασπιζόμαστε τις πιο μικρές επιχειρήσεις που είναι και οι πιο αδύναμες. Θα θέλαμε να εισακούστούμε και θα ήθελα να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά μέχρι ότου εξευρεθεί μία τελική λύση. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε. Ο κύριος Χεντομένης έχει το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής. Η αναφορά 500 κάθετος 2010 υποβλήθηκε από τον δόκταρα Ντεμπόνης εξ ονόματος της ΑΝΛΑΚ της ε, ε, Ένωσης Εκτροφέων Κουνελιών. Στην ε, αναφορά αυτή ότι ο τομέας εκτροφής του, των κουνελιών στην Ιταλία γνωρίζει μία βαθύτατη ε, κρίση εδώ και τρία χρόνια και παρά την εσωτερική κατανάλωση, η οποία είναι πολύ υψηλή, η Άνλακ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Από το 2007 η εκτροφής κουνελιών παρήγαγαν 93.000 ε, τόνους, δηλαδή 67 εκατομμύρια κεφαλές και ήταν η ε, δεύτερη ε, εκτροφές του κόσμου μετά από την Κίνα. Η Άνλακ, όπως είπε και ο κύριος Ντεμπόνης, επέσυρε την προσοχή της Ιταλικής κυβέρνησης στην κατάσταση κρίσης του τομέα, αλλά η Ιταλική κυβέρνηση δεν έχει προσδώσει τους κατάλληλους πόρους για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση αγοράς. Όπως ε, τόνισε και ο αναφέρον, η ΑΝΛΑΚ πρόσφατα υπέβαλε ε, δύο αναφορές δυνάμει του άρθρου 101 και 102 για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν κάνω λάθος, στις 10 ε, Σεπτεμβρίου ε, απορρίφθηκε η πρώτη καταγγελία, ενώ η δεύτερη εξετάζεται από την ε, Εθνική Αρχή, Εθνική Εγγυητική Αρχή. Ε, χτες ε, μίλησα με την αρμόδια αρχή η οποία μου είπε ότι εξετάζει με ενδιαφέρον τα έγγραφα αυτά της ANLAC. και νομίζω ότι στις 18-20 ε, Νοεμβρίου, δύο εβδομάδες δηλαδή πριν, συντάχθηκε ένα λεπτομεριακό ε, μνημόνιο 60 σελίδων που διάβασα με μεγάλο ενδιαφέρον διότι τότε μας ε, διαβιβάστηκε. Θα ήθελα να πω ότι η Unlock δεν έχει προβεί σε μια καταγγελία προς ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δυνάμει των Άρθρων 101 και 102. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω αυτά τα οποία ε, έχω καταγράψει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στο υπάρχον σύστημα. Το υπάρχον σύστημα βασίζεται στη, στη απόφαση του Συμβουλίου του 2003 και στο διάταγμα της αρχής εγγύησης του ανταγωνισμού. Μιλάμε για ένα παράλληλο σύστημα αρμοδιοτήτων όπου η εγγυητική αρχή ανταγωνισμού και η Επιτροπή μπορούν να εφαρμόσουν τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης περί λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα δίκτυο που λειτουργεί για το δημόσιο συμφέρον ο κανονισμός 1 κάθετος 2003 ε, και η ανακοίνωση της Επιτροπής έχουν ως στόχο ε, τον επιμερισμό, σωστό επιμερισμό εργασίας μεταξύ κομισιών και εθνικών αρχών ανταγωνισμού. Αυτό το σύστημα ορίζει ότι για να εφαρμοστούν τα άρθρα 101 και 102 θα πρέπει η Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβούν σε μία ανακοίνωση επί του θέματος. Τη στιγμή που υπάρξει επίσημη καταγγελία, τότε η πρώτη αρμόδια αρχή κρατά αυτή, ασχολείται με αυτή την ε, υπόθεση και δεν γίνεται επανακατανομή εκτός και αν υπάρχει μία άλλη αρχή που βρίσκεται σε καταλληλότερη θέση να κρίνει ή να παρέμβει. Και τότε δεν υπάρχει θέμα διακριτικής ευχέρειας. Όταν μία αρχή ε, μπορεί να ε, παρέμβει, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη εάν πληρούνται συγκεκριμένοι όροι. Εάν υπάρχουν άμεσες συνέπειες, απρόβλεπτες συνέπειες στην εθνική επικράτεια και να δούμε κατά πόσο ε, υπάρχουν στοιχεία που απορρέουν από τα συγκεκριμένα δεδομένα. Τότε ξεκινά η διαδικασία παραβίασης και θα πρέπει να δοθεί, να εκδοθεί ένα διάταγμα παύσης εργασιών, διακόπτει ο μιλητής, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με τα μικρόφωνα. Άρα, όπως έλεγα, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά τρεις όροι. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να δράσουν με βάση την, ε, μια πρακτική που αντιβαίνει στις αρχές του ανταγωνισμού και με βάση τις, τις πάγιες πρακτικές στην εθνική επικράτεια. Δεύτερον, θα πρέπει να παρέμβει για να θέσει τέλος στην παραβίαση αυτή, επιβάλλοντας κυρώσεις στους αντιβαίνοντες και να συλλέξει τα στοιχεία τα οποία συντείνουν υπέρ της παραβίασης. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί τέλος στην κατακριτέα αυτή πρακτική και να συλλεχθούν τα αποδεικτικά στοιχεία έτσι ώστε να αποδειχτεί αυτή η παραβατική ε, πράξη. Στην περίπτωση της Άνλακ αυτά τα τρία κριτήρια πληρούνται όσον αφορά τις Ιταλικές αρχές. Θα πρέπει λοιπόν να θεωρήσουμε ότι οι Ιταλικές αρχές ανταγωνισμού είναι στην ε, σωστή και κατάλληλη θέση για να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα. Εξάλλου, όπως προείπα, είμαστε σε επαφή με τις Ιταλικές αρχές και οι Ιταλικές αρχές εξετάζουν το θέμα. Άρα, η Επιτροπή ε, δυνάμη του ρυθμιστικού πλαισίου δεν μπορεί να παρέμβει έναντι αυτών των πρακτικών. Έναντι των επιχειρήσεων, όπως καταγγέλει η Άνλακ. Βεβαίως, η Επιτροπή θα συνεργάζεται με τις ταλικές αρχές ανταγωνισμού, έτσι ώστε να έχουμε μία σωστή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού με βάση τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνάμει των άρθρων 101 και 102. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελα να παρέμβει κάποιος συνάδελφος. Oui. Je... Θα ήθελα απλώ για το θέμα αυτό να πω ότι ναι, πρέπει να μην ανοιχτή η αναφορά, φαντάζομαι, αφού επισημένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σκοπεύει να συνεργαστεί με την Ιταλία. Φαντάζομαι ότι η Ένωση θα ήθελε να δει επιτάχυνση τη διαδικασία. αφού είναι παραγωγή. Έτσι δεν είναι και άρα έχουν οικονομική ζημιά από την καθυστέρηση. Μπορούμε να αισθήσουμε επιτάχυνση αυτής της μελέτης από πλευρά τη Ιταλία. Εγώ αυτό θα προτείνω. Και να μείνει ανοιχτή η αναφορά για να δούμε και τη συνεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πράξη. Συμφωνώ με τη συνάδελφη. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, γι' αυτό υπό το φως αυτών που μας προείπε ο εκπρόσωπος Επιτροπής θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, διαδικασία αυτή καταγγελίας και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού. Άρα θα πρέπει να προωθηθεί η συνεργασία αυτή όπως προβλέπει η Επιτροπή και νομίζω ότι μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό το δίκτυο που ελέγχει τον ανταγωνισμό και τις συνθήκες ανταγωνισμού. Μπορούμε να αποστείλουμε ένα υπόμνημα ως ε, Επιτροπή για να ε, μάθουμε για την εξέλιξη της διαδικασίας διότι Φυσικά δεν θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση από την Εκτελεστική Επιτροπή, όμως ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κατά πόσο θα πρέπει να προωθήσουμε μια διαδικασία διερεύνησης με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα πρέπει να ζητήσουμε μια επιτάχυνση της διαδικασίας, διότι αν υπάρχει παραβίαση του ρυθμιστικού πλαισίου θα πρέπει να παρέμβουμε εγκαίρως. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τις Ιταλικές Αρχές να επιταχύνουν αυτή τη διαδικασία επαλήθευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Ιταλικές Αρχές ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα και μίλησαν και ενέκριναν μάλλον τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου χωρίς όμως να φτάσουν σε ένα τελικό συμπέρασμα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς ως Επιτροπή Αναφορών να ζητήσουμε επιτάχυνση των διαδικασιών από τις Ιταλικές Αρχές. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Συμφωνεί και η κυρία Γκρουνή. Αφήνουμε ανοιχτή λοιπόν αυτή την αναφορά. Περνάμε στο επόμενο θέμα που αφορά το σημείο 9 ο αναφέρον δεν είναι παρόν, άρα δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Η αναφορά αφορά τον κύριο Λοράν Ερμουά, εξ ονόματος της Ένωσης για την Προωσία των Δικαιωμάτων των Ειδικευόμενων Ιατρών σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των Ειδικευόμενων Ιατρών στο Βέλγιο. Έχετε το λόγο. Yes, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μια αναφορά για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει ανακοίνωση τον Οκτώβριο του 2008 και τον Οκτώβριο του 2009 στην ε, Επιτροπή σας ε, και ευχαριστώ να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις. Η αναφορά αφορά την αδυναμία των βελγικών αρχών να μεταγράψουν την οδηγία για το χρόνο εργασίας ε, σε σχέση με τους χρόνους εργασίας ε, των ε, ειδικευομένων γιατρών σε δημόσια νοσοκομεία στο Βέλγιο. Ο αναφέρον ε, σωστά έθεσε το θέμα λέγοντας ότι συνεπώς ε, δεν υπήρχε όριο στο χρόνο εργασίας ε, για τους ειδικευόμενους ιατρούς στα βελγικά νημόσια νοσοκομεία και συνεπώς δεν θα μπορούσαν, δεν θα μπορούσαν να καλούνται να δουλεύουν ε, για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, μέχρι και 80 ώρες την εβδομάδα. Κάνουν επίσης συναπτές βάρδιες, ε, οι οποίες φτάνουν μέχρι και τις 36 ώρες, χωρίς διάλειμμα, κάτι το οποίο αντίκειται στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τις βελγικές αρχές ε, προκειμένου να ενημερωθεί για τη θέση τους. Ε, μεταγράφηκε τελικά ε, η οδηγία από τις βελγικές αρχές, όμως ε, το μέτρο μεταγραφής στη συνέχεια ακυρώθηκε για λόγους διαδικασίας από ένα διάταγμα του Συμβουλίου Επικρατείας και συνεπώς δεν μεταγράφηκε όντως τελικά η οδηγία. Στην τελευταία μας ανακοίνωση ε, αποστήλαμε επιστολή στις βελγικές αρχές το Νοέμβριο του 2009 σε σχέση με τη συμμόρφωσή τους ε, με την οδηγία επί πολλών θεμάτων, οι βελγικές αρχές ε, στη ε, συνέχεια προετοίμασαν ένα νέο νόμο για τη μεταγραφή της οδηγίας για τις συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων. Παρακολουθήσαμε την πρόοδο του νόμου, παρουσιάστηκε το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, αλλά λόγω της τρέχουσας πολιτικής κατάστασης στο Βέλγιο μετά από τις τελευταίες εκλογές υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις με την οροστικοποίηση και την έγκριση του μέτρου, αλλά ενημερωθήκαμε ότι εγκρίθηκε από ε, το ε, Κοινοβούλιο, έχει υποβληθεί ε, στην Γερουσία και, περιμέν, και αναμένεται η έγκρισή του μέχρι το τέλος της χρονιάς ή το πολύ στις αρχές της επόμενης χρονιάς. Ενημερωθήκαμε από τις βελγικές αρχές ε, ότι υπήρξαν τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των νοσοκομείων, των ειδικευμένων ε, ιατρών ε, και τη κυβέρνησης ε, καλύπτονται βέβαια και άλλες ομάδες όπως ε, οι ιατροί, οι ε, δικαιωμένοι οδοντίατροι ή κτηνίατροι που είχαν αποκλειστεί από την προηγούμενη μεταγραφή της οδηγίας. Η έκβαση της μετάφρασης, της μεταγραφής, συγγνώμη, είναι ότι η κατάσταση θα διορθωθεί σε σημαντικό βαθμό με τη σωστή εφαρμογή της ε, των τελευταίων μέτρων ε, θα υπάρξει νέα νομοθεσία η οποία θα θέτει ένα όριο στον μέσο όρο εβδομαδιαίας εργασίας των ειδικευμένων γιατρών και θα εξασφαλίζει ότι ότι θα ε, έχουν ε, χρόνο ανάπαυσης ε, ως αντιστάθμιση στις υπερορίες ή στις βάρδιες, γιατί δεν ζητήθηκε opt-out βάσει του άρθρου 32 της οδηγίας, γιατί βάσει του οποίου θα μπορούσε ένας ειδικευμένος, ειδικευόμενος γιατρός να ζητήσει να υπερβεί το όριο του χρόνου εργασίας προβλέπεται από την οδηγία, κάτι το οποίο επιτρέπεται φυσικά από την οδηγία. Υπάρχει όμως ένα όριο στον αριθμό των επιπλέον ωρών εργασίας. Ε, είναι ένα συνολικό όριο 12 επιπλέον ωρών ανά εβδομάδα. Και βέβαια ε, υπάρχουν ε, κάποιοι όροι προστασίας για τη ε, χρήση του opt-out, οι οποίοι επίσης ε, μετεγράφησαν. Θα δούμε λοιπόν όταν θα αρχίσει να ισχύει το μέτρο πώς εφαρμόζεται, αλλά κατά την άποψή μας είναι ικανοποιητική η ανταπόκριση των βελγικών αρχών. Υπάρχουν συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο. Η ναι, κυρία Γκρουινή. Θα ήθελα απλώς να πω ότι δεν θα πρέπει να ε, κλείσουμε την υπόθεση, ούτως, ε, την αναφορά της αυτήν την υπόθεση, να περιμένουμε να δούμε την ε, μεταφορά στο βελγικό δίκαιο. Και πάλι να δούμε αν τώρα αυτή τη φορά εφηγραμμίζονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο κατά την μεταφορά της οδηγίας. Δεν υπάρχουν δηλαδή προβλήματα να περιμένουμε την μεταφορά πριν να κλείσει η αναφορά ο κύριος Μπροστινάρου και εγώ συμφωνώ απολύτως με την ε, ιδέα της συναδέλφου να παραμείνει ανοιχτό, ανοιχτή αναφορά μέχρι να υλοποιηθεί από την εθελεστική εξουσία του Βελγίου. Όποια είναι αυτή τέλος πάντων. Όποια κυβέρνηση. Και επίσης το αποτέλεσμα της ε, αναφοράς επιβεβαιώνει τη βούληση της Επιτροπής των Αναφορών και την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής των Αναφορών. Μπορεί να επιφέρει ακόμη και τροποποίηση της νομοθεσίας σε ένα κράτος μέλος, εάν αυτή η νομοθεσία παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ή αν μια σχετική απόφαση κάποιες αρχής αρμόδια σημεί ε, παραβιάζει το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστό να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, διότι η απάντηση της Επιτροπής μας προτρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία επαλήθευσης από πλευράς εθνικών αρχών της, του κοινοτικού ρυθμιστικού πλαισίου. Είμαστε σε επαφή λοιπόν με την επαφή για να, ε, ε, σε επαφή με την Επιτροπή για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Σημείο 10. Αναφορά της Παλίνας Ικός Καράμπεκ, πολωνική σταγένεια σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης των πολωνών γιατρών που εργάζονται στο μέα της δημόσιας υγείας. Και Κρίστοφ Μπούκελ αναφορά επίσης πολεμικής εχαγένειας του κ. Μπούκελ, εξ ονόματος της ΟΖΛ της Εθνικής Συνδικαλιστικής Ένωσης Ιατρών όπου, η οποία συνοδεύεται από 6.770 υπογραφές. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Yes, thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε δει να κάνουμε μια, άλλη, μια ακόμη αναφορά που σημειώθηκε σημαντική πρόοδος από τη στιγμή που αρχικά είχαν υποβληθεί οι αναφορές. Ε, λίγο πολύ καλύπτουν το ίδιο πεδίο, δηλαδή έχουν να κάνουν με την ευθυγράμμιση πολωνικής νομοθεσίας στην ε, παροχή υπηρεσιών υγεία υγείας ε, στην οδηγία πλαίσιο και συγκεκριμένα και επίσης την ομολογία του, δικαστηρίου ως προς την, νομοθεσία Γέγκερ, την ομολογία Γέγκερ για τον τρόπο με τον οποίο η πολωνική νομοθεσία αντιμετωπίζει τον χρόνο ε, εργασίας και, και εφημερίας. Είχε σημειωθεί λοιπόν αρχικά ότι ήταν προβληματική, δεν ήταν αρκετά ευθυγραμμισμένη πολωνική νομοθεσία στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ωστόσο οι εθνικέ αρχέ πρέπει σε σημαντικέ ε, τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία που ετέθησαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2008 ύστερα από αρκετές ε, δικαστικές αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων της Πολωνική που επέμειναν στην αρχική, αρχικά, εξ αρχή, μάλλον, στην ορθή εφαρμογή των ε, νόμων. Ύστερα λοιπόν από τις σχετικές ε, τροποποίησει. πρώτον ο, χώρος εφημερία, ο χρόνος εφημερίας, το χρόνο εργασίας υπολογίζεται σωστά, με βάση και τις αποφάσεις Διακού και δεύτερον ορίζεται όριο, το όριο 48 ετο, ε, ωρών την εβδομάδα ε, για την ευημερία των ε, ιατρών στην Πολωνία. Τρίτον, οι ιατροί παίρνουν τώρα ρεπό στο χρονικό πλαίσιο που έχει ζητήσει και επιβάλλει η απόφαση Διέγου, όπου προσωρινά υπάρχει καθυστέρηση στην αναπλήρωση αυτή, στην ανάβαυση και τέταρτον ε, γίνονται από ό,τι μαθαίνουμε ε, έλεγχοι, έγιναν ιδιαίτερα το 2008 εκταμένη έλεγχοι από την ε, επιθεώρηση εργασίας στα νοσοκομεία για να βεβαιωθεί ότι όντως πληρούνται αυτές οι προδιαγραφές της νομοθεσίας. Για δε τη δεύτερη αναφορά. όπου αναφερόμενος είχε ξεκινήσει ανταλλαγή επιστολών με την Επιτροπή για το θέμα που τον απασχολούσε. Επαληθεύσαμε λεπτομερώς την εφαρμογή στην πράξη των ε, σχετικών διατάξεων του πολωνικού δικαίου. Πρέπει να πω ότι κάποιες από τις παρατηρήσεις των αναφορών ε, είναι εκτός του πεδίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου, κυρίως όσον αφορά τις παρατηρήσεις τους για την ε, επαρκή αμοιβή των ε, ιατρών και των τιμολογίων για τις αμοιβέ των γιατρών. Οι άλλες παρατηρήσεις σχετικές ε, με τον υπολογισμό του χρόνου εφημερίας για την κοινωνική ασφάλιση των ιατρών. Αυτά τα τρία θέματα είναι έξω από το ευρωπαϊκό δίκαιο και άρα μπορούν να ρυθμιστούν αποκλειστικά και μόνο από το εθνικό. Σε κάποια σημεία στα οποία έχουμε από την προηγούμενη μας απάντηση εκφράσει κάποιες ανησυχίες και είχαμε πει ότι θα θέλαμε πριν να επανέλθουμε στην Επιτροπή των Αναφορών να δούμε κάποιες απαντήσεις, ήταν τα εξή. Το πρώτο, το οποίο θεώρησε μάλλον σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν ένα ζήτημα το οποίο έθεσε ο δεύτερος αναφερόμενος στην ε, επιστολή του στην Επιτροπή Αναφορών το Μάρτιο του 2008 όπου καταγράφονταν επεισόδια σε ένα συγκεκριμένο ε, νοσοκομείο της ε, Πολωνίας όπου είχε ζητηθεί από γιατρούς να μείνουν στη δουλειά περισσότερο από τους 48 τα δυνάμει ενός opt-out που είχε στην περίοδο εκείνη ακόμη η Πολωνία, είχαν αρνηθεί οι ιατροί και στη συνέχεια, από ό,τι είπε ο αναφερόμενο, απειλήθηκαν ότι θα κλείσει το σχετικό, η σχετική κλινική του νοσοκομείου και ότι θα έχαναν τη δουλειά του. Στη νομοθεσία λοιπόν προβλέπεται ότι εφόσον δεχθεί να εργαστεί άνω του 48 ωραίου ο ιατρός θα πρέπει η συνένεσή του να είναι ελεύθερη και χωρίς η πίεση, χωρίς να έχει υποστεί αυτός η πίεση. Και ως εκ τούτου εμείς αποστήλαμε επιστολή μόλις ενημερωθήκαμε για την ε, περίπτωση αυτή και στις εθνικές αρχές αλλά και στις ε, οργανώσεις των αφαιρωμένων ζητώντας διεξοδική ενημέρωση και από τις δύο πλευρές για το τι ακριβώς είχε συμβεί. Και οι δύο πλευρές μας έστειλαν λεπτομερή στοιχεία για τα επεισόδια αυτά. Συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ερμηνευθούν τα επεισόδια αυτά και ιδιαίτερα με την δεύτερη πλευρά, δηλαδή την οργάνωση των αναφερομένων. Η Επιτροπή έχει κάποιες ανησυχίες για τις δράσεις που φαίνεται πως ανέλαβαν κάποιες δημόσιες αρχές στο θέμα αυτό. Inspections uh, Πάντως φαίνεται πως οι επιθεωρητές υγείας, η εργασίας μάλλον, που έλεγξαν εάν οι εμπλεκόμενοι γιατροί υπέστησαν κάποιες κυρώσεις όταν δεν δέχθηκαν να ξεπεράσουν τα οκτάρο. Και φαίνεται ότι δεν υπήρξε αντίρρηση ή ένσταση από πλευρά των εμπλεκομένων γιατρών στην απόφαση αυτή. Ε, έτσι λοιπόν προκύπτει πως δεν υπάρχει λόγος η Επιτροπή να αναλάβει αδίποτε δράση ως προς Κυρώσει κυρώσεις εις βάρος των ιατρών αυτών για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η επιστολή που αποστήλαμε στις αρχές φαίνεται πως βοήθησε και διαλύθηκαν κάπω την κατάσταση για όλες τις πλευρές και πιστεύουμε ότι δεδομένου της έκβαση αυτής δεν είναι εφικτό ή χρήσιμο λυσιτελές αυτή τη στιγμή να αναλάβουμε περαιτέρω δράση. Φαίνεται ότι επαναπροσλήφθηκαν αυτοί οι ιατροί εντωμεταξύ και ότι δεν υπήρξαν άλλα τέτοια επεισόδια στο ίδιο νοσοκομείο. Η επιστολή των αφαιρωμένων ε, επιστήμων και κάποια άλλα σημεία που γίνουν ανησυχία και που θέλαμε να διερευνήσουμε περισσότερο. Φαίνεται ότι Υπάρχει η πρακτική να προσλαμβάνονται με πολλαπλέ συμβάσει, δηλαδή διαφορετικέ ώρε εργασία με διαφορετικέ συμβάσει οι ιατροί. Αποτέλεσμα είναι να ξεπερνούν του 48 ώρου. Από την ε, διερεύνηση της υπόθεσης φαίνεται πως υπάρχουν διάφορες πρακτικές εδώ, περίπλοκες. Σε ορισμένε περιπτώσεις οι συμβάσεις φαίνεται να συνάπτονται ως συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και όχι έργου. Και είναι πολύ δύσκολο να διευκρινιστεί εάν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογή της οδηγίας αυτής για το χρόνο εργασίας. Όταν έχουν πάνω από έναν εργοδότη, αντισυμβαλόμενο ή εργαζόμενο, υπάρχει ζήτημα, και αυτό συστήθηκε διεξοδικά κατά τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο, και πιστεύουμε ότι και πάλι θα συζητηθεί στη νέα αναθεώρηση το 2011 ο τρόπος υπαγωγής αυτών των συμβάσεων στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε σαφείς αποφάσεις για το ευρωπαϊκό δίκαιο έτσι ώστε κατά πιο αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίζονται στο μέλλον τέτοιου προβλήματα. Και εν τέλει, λαμβανομένων υπόψη και των συζητήσεων που μπορέσαμε να αναπτύξουμε μέσω και άλλων διάβλων με τον αναφερόμενο και των ερευνών μας μέχρι σήμερα. Φρονούμε πως όπως έχει η κατάσταση η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει περαιτέρω λυσιτελή δράση και όταν σε κάποια περίπτωση επρόκειπταν δυσκολίες στην ερμηνεία του εθνικού δικαίου θεωρήσαμε ότι ήταν σκοπιμότερο να διευκρινιστούν οι διατάξει τη οδηγία στην προσοχή αναθεώρηση που αναμένεται το 2011. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να παρέμουν, κυρία Γκρινή αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει περισσότερα και επειδή υπήρξαν και υπήρξε και θετική ανταπόκριση από πλευράς ε, ε, του κράτους μέλους, μήπως μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Και αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα μπορούν να υποβάλουν νέα αναφορά. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να κλείσουμε την αναφορά αυτή. Κύριε Μποστινάρου. Και εγώ συμφωνώ να το κλείσουμε εδώ το θέμα της αναφοράς αυτής και διαπιστώνω ότι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένει ελαφρώς αμφίσιμη. Και αυτό μας δημιουργεί άγχος. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη που πρέπει να διερευνήσει Είτε πρόκειται για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είτε όχι. Αν υπάρχει παραβίαση, παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, πρέπει να καταλήξουμε σε μια διαδικασία κυρώσεων, αν χρειάζεται, ε, για να, ή να βελτιώσουμε την εθνική νομοθεσία για να συμμορφωθεί η νομοθεσία αυτή με το ε, ευρωπαϊκό δίκαιο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή μας λέτε περίπου ναι και όχι για το θέμα αυτό. Είναι δύσκολο και για μας τους ευρωβουλευτές να, κρίνουμε την κατάσταση, αλλά συμφωνώ με την κυρία Γκρινή να κλείσει εδώ αυτό το θέμα. αλλά ίσως θα έπρεπε στο μέλλον να αποφεύγουμε τις πολύ αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Θα πρέπει να πω ότι δεν συμμερίζομαι αυτή την πρόταση, αλλά θα δεχτώ τη θέση της πλειοψηφίας. Διότι η Επιτροπή δήλωσε ότι υπάρχει παραβίαση και μιλά για μια διαδικασία παλήθευσης και κοινοποίησης της παραβίασης προς εθνικές αρχές. Θα πρέπει να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία σε αυτή την περίπτωση. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε ότι στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, κατά πόσο στην περίπτωση μη συμμόρφωσης θα έπρεπε να δράσουμε έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να είναι αποκλειστικά υπεύθυνες. Άρα, σε αυτή την περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να κρίνει μόνο εάν έχουν συμμορφωθεί οι εθνικές αρχές. Αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μια συνεργασία με τους ε, πολίτες και να δούμε κατά πόσο η προσαρμογή συντελείται όπως πρέπει. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας διευκρινίσει η Επιτροπή. Υπάρχουν σημεία όπου υπάρχει αμφισημία σύμφωνα με την Επίτροπη και θα πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξει μελλοντικά η ίδια η οδηγία. Δεν έχω κατανοήσει αυτή την τελευταία διατύπωση γιατί πρόκειται σαν να είναι, μια, είναι σαν μια έκκληση για να αλλάξει το κανονιστικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή. Ναι, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, σωστά έπρεπε να είχα εξηγήσει λίγο την ιστορία της υπόθεσης. Ε, υπήρχε μία πρόταση από το 2004 στο 2009 για την τροποποίηση της ε, οδηγίας για το χρόνο εργασίας για πάρα πολλά ζητήματα και Παρά το γεγονό ότι έγιναν πολλέ αναγνώσει και διαδικασία συνδιαλλαγή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν συμφώνησαν ε, για τι αλλαγέ που έπρεπε να γίνουν και συνεπώ κατέπεσε η πρόταση. Indeed, Mr. the rapporteur. Ο κύριος ε, Τσίρκας που είναι ε, ο εισηγητής το γνωρίζει. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ο κύριος Μπαρόσο, ανακοίνωσε στο Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο ότι θα προτείνει αναθεώρηση της οδηγίας για το χρόνο εργασίας και ότι θα γίνει και διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, όπως επιζητά και η συνθήκη. Επίσης θα γίνει μια λεπτομερής μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου. Αυτή τη στιγμή ε, γίνεται διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ε, και διενεργούνται και οι μελέτες αξιολόγησης αντικτύπου. Αποστήλαμε το Μάρτιο το πρώτο έγγραφο διαβούλευσης ε, και το δεύτερο αναμένεται να εγκριθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Οπότε πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας ε, θα προταθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, την επόμενη χρονιά, γιατί πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα διάφορα στάδια διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ποιο θα είναι το πεδίο εφαρμογής της νέας αυτής πρότασης και δεν υπάρχει και απόφαση καμία για το περιεχόμενο της συγκεκριμένης αναθεώρησης και περιμένουμε να ολοκληρωθούν και να ολοκληρωθεί το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Πριν από τα Χριστούγεννα θα αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βέβαια και στο Συμβούλιο και στους κοινωνικούς εταίρους, διάφορες μέθοδοι ε, αναθεώρησης, πιθανές μέθοδοι ανανεώρησης. Τώρα, σχετικά με το αν υπάρχει συμμόρφωση ή όχι. Συγγνώμη, εγώ δεν ήθελα να δημιουργηθεί οποιαδήποτε αμφιβολία σε σχέση με αυτά που είπα. Πρόκειται για έναν ε, τομέα που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας χρόνου εργασίας στα νοσοκομεία ε, σε σχέση με τους χρόνους ε, εφημερίας. Αυτές είναι οι δυσκολότερες, οι πιο προβλημα... οι δυσκολότεροι οι πιο προβληματικοί τομείς εφαρμογής της συγκεκριμένη οδηγίας και ήμασταν πολύ προσεκτικοί. Αυτή τη στιγμή γίνονται αλλαγές στην εθνική νομοθεσία Γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές θέλουμε να επανέλθουμε σε επιπρόσθετα ε, σημεία ε, από το Δεκέμβριο του 2009 και μετά. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των ε, ιατρών για τους οποίους υπάρχουν ισχυρισμοί ότι υπέστησαν πίεση να συγκατατεθούν ε, για το opt-out που προβλέπει η οδηγία και συνεπώς να δουλέψουν περισσότερο, είναι κάτι το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό γιατί είναι παραβίαση του θεμελιώδους, ε, της θεμελιώδους αρχής ε, ότι δεν πρέπει να υποχρεώνεται κανείς να δουλεύει πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα δεν ε, υπήρξαν ενδείξεις ε, από τους αναφέροντες ε, ότι υπήρξαν προβλήματα και έρευνές μας δεν κατέδειξαν κάτι τέτοιο. Οπότε πραγματικά αυτός ο ισχυρισμός τότε μας είχε ανησυχήσει πάρα πολύ, όμως δεν έχουμε ενδείξεις ότι επαναλήφθηκε το φαινόμενο και ούτε ε, και λάβαμε ενημέρωση από τους αναφέροντες ότι είχαν προσληφθεί όλοι ε, οι ιατροί και συνεπώς δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν βλέπουμε λοιπόν Πώ παραβίαση τη κοινωνική νομοθεσίας. Σε σχέση τώρα με, τα, με τους ιατρούς ε, που έχουν πολλαπλές συμβάσει με το ίδιο νοσοκομείο και αυτό σημαίνει ότι δουλεύουν περισσότερο από 48 ώρες ε, την εβδομάδα. Από τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας ε, φαίνεται ότι αυτό γίνεται μέσω συμβάσεων που δεν είναι συμβάσεις εργασίας Δηλαδή, εργάζεται ως υπάλληλο ο γιατρός για το νοσοκομείο, αλλά, επιπλέον, αλλά παρέχει και επιπλέον ε, ε, υπηρεσίες ως εξωτερικός ιατρός, για να το πω έτσι, κάτι το οποίο επιτρέπεται. Δεν μας αρέσει βέβαια ιδιαίτερα αυτή η πρακτική, αλλά κατά αναλογία με το opt-out δεν μου είναι πάρα πολύ σαφέ κατά πόσο αυτό είναι παραβίαση της οδηγίας αν ο γιατρό λαμβάνει ελεύθερη απόφαση να δουλέψει επιπλέον ώρες. Άρα θα προτιμούσαμε να το εξετάσουμε αυτό με διευκρίνηση των διατάξεων της ίδιας της οδηγίας, των διατάξεων που δεν είναι πάρα πολύ σαφή σε σχέση με την εφαρμογή ε, της οδηγίας στην περίπτωση των πολλαπλών συμβάσεων και, και βέβαια μέσω επαφών με τις εθνικές αρχές να μπορούμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να οριοθετήσουμε περισσότερο συμβάσεις ε, οι οποίες ε, είναι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και που λαμβάνονται ελεύθερα ως, απόφαση, ε, ελεύθερη απόφαση από τους ιατρούς ή εμπίπτουν στο δίκαιο των συμβάσεων εργασία με το νοσοκομείο. Ε, πρέπει να υπάρχει και συνεργασία με τους μηχανισμούς, για, τους, για τους μηχανισμούς επιβολής και γι' αυτό ακριβώς ζητούμε τη συνεργασία των κρατών μελών προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει επίσης ένα ακόμη ζήτημα και αφορά ε, που αφορά τη συμμόρφωση με την οδηγία, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα. Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή ποια είναι τα όρια εφαρμογής της οδηγίας. Δεν είμαι ούτε εγώ απολύτως ικανοποιημένη, αλλά υπάρχει μια έλλειψη ε, ε, σαφήνεια σε σχέση με αυτό. Σας ευχαριστώ για τη δεύτερη αυτή παρέμβαση. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, τότε θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Κυρία Γκρουνή. Κοιτάξτε, εγώ προτείνω να κλείσουμε τη συγκεκριμένη αναφορά διότι δεν υπάρχει απόδειξη ότι το κράτος μέλος ή το νοσοκομείο ε, δεν έχει συμμορφωθεί με την οδηγία και δεν μπορούμε να ε, την αφήσουμε ανοιχτή περιμένοντας τι θα γίνει με την αναθεώρηση της οδηγίας. Μπορεί ας πούμε να δεχθούμε ε, σε μεταγενέστερο στάδιο μία αναφορά αν παραβιάζεται το κοινοτικό δίκαιο στο μέλλον. Για μένα λοιπόν πρέπει να κλείσει η συγκεκριμένη αναφορά. Όπως σας είπα υπάρχει, έχει διαμορφωθεί μία πλειοψηφία άρα δεν υπάρχει καμία Μία αμφιβολία σε σχέση με το κλείσιμο αυτής της αναφοράς. Μπορούμε να προχωρήσουμε με την υπαριθμόν 11 του Μάρκ Σάζιεκ που είναι παρόν, άρα του δίνω το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, μέλη τη Επιτροπή των Αναφορών. Σα ευχαριστώ εκ μέρου όλων των εργαζομένων στα ασθενοφόρα ε, μισθωτών και ιδιωτών από τη Γαλλία που ήρθαν εδώ να αναφερθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και θα ήθελα επί τη ευκαιρία να σας εκθέσω τις διεκδικήσεις μας. Ο χρόνος εργασίας των εργαζομένων, των μισθωτών στα ασθενοφόρα υπόκειται σε ένα σύστημα ισοτιμίας που θεσπίστηκε με μια συμφωνία πλαίσιο το Μάιο του 2000 έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη και η περίοδοι αδράνειας ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εφημερίας, ανάπαυσης γευμάτων, διακοπών και οι εναλλαγές στην ένταση της αστεριότητας. Έτσι λοιπόν ε, δεν λαμβάνονται υπόψη ε, ή καλύτερα δεν αξιολογούνται επαρκώς η διάρκεια παρουσίας των χρόνο εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, κατά καταδίκασε το 2005 ε, κατήγγειλε μάλλον την, το διάταγμα 2001-1381 το οποίο ήταν αντίθετο με την κοινωτική οδηγία το οποίο δεν αφορούσε τους εργαζόμενους στην, ε, ε, χώρο των ασθενοφόρων αλλά το οποίο σας έχουμε συ, το οποίο έχουμε περιλάβει στην αναφορά μας. Το διάταγμα 2009-32 της 9ης Ιανουαρίου 2009 κατήργησε και αντικατέστησε το διάταγμα 679-2009 του οποίου ζητούσαμε και εμεί με την αναφορά μας την κατάργηση πριν όμως διατηρούνται ορισμένε ε, ισοτιμίες όσον αφορά το σύστημα υπολογισμού του χρόνου εργασίας με έναν ε, συντελεστή 80 με 90% για όλους τους εργαζομένους στα αστυνοφόρα και λεσίδε 75% για τι εφημερίε. Όμω εμεί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια είναι τα ωράρια εργασία μα εκ των προτέρων και είμαστε πάντα στη διάθεση τη επιχείρηση για την οποία εργαζόμαστε, διότι δεν μπορεί να προβλεφθεί πόση δουλειά θα προκύψει κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν είναι ε, ουτοπικό να πιστεύει κανεί ότι ε, ο μισθωτό στα χώρο των ασθενοφόρων μπορεί να διαθέσει ελεύθερα το χρόνο του κατά τη διάρκεια της αδράνειας γιατί του πάντα έχει και δουλειά να κάνει όπως ε, να ε, ενημερωθεί περισσότερο, να ε, αποκαταστήσει το υλικό του, να το απολυμάνει κτλ. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ειδικέ παρεκκλήσεις σε σχέση με το επάγγελμά μας. Υπάρχουν διακοπές οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη σε περίπτωση απρόβλεπτων αποστολών. Υπάρχει καθυστέρηση εναλλαγή αλλαγή μάλλον του χρόνου ε, των γευμάτων, των καθημερινών ωρών εργασίας που μπορεί να φτάσουμε και 15 την ημέρα, τη ημερήσιας ανάπαυση κτλ. Αυτές όλες οι παρεκκλήσεις λοιπόν ε, συγκεντρώνονται, συσσωρεύονται εις φάρος του ε, εργαζομένου, δυστυχώς δεν υπολογίζονται αυτά τα δυσάρεστα χαρακτηριστικά της δουλειάς μας ε, και, και υπολογίζεται μόνο η περίοδος αδράνειας ως χρόνος εργασίας. Είναι άδικο λοιπόν να μην ε, να μην αμείβονται με τον ίδιο τρόπο οι εφημερίες μας λόγω των ε, και αυτό το ζητούμε λόγω των διαταραχών που μπορεί να καλέσουν στην κοινωνική και οικογενειακή ζωή μας αλλά και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στην υγεία μας. Έτσι λοιπόν ζητούμε να αλλάξουν αυτοί οι συντελεστές, να καταργηθούν αυτοί οι συντελεστές και να καταργηθεί και το διάταγμα 2009-32 της 9ης Ιανουαρίου 2009 που τους επιβάλλει τους συντελεστές αυτές. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο έχει και πάλι η Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μία αναφορά ε, στην οποία απάντησε εγγράφος με πολύ λεπτομέρεια τον Οκτώβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε ζητήσαμε περαιτέρω διευκρινήσεις ε, σε σχέση με τα ε, γεγονότα και ο αναφέρον ε, παρήχε κάποιες διευκρινήσεις ε, σε σχέση με την αλλαγή της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. Πρόκειται για μια, ένα πολύ τεχνικό τομέα του χρόνου εργασίας και θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι διακυβεύεται και τι έχει αναφερθεί στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το βασικό ζήτημα είναι ο υπολογισμός ε, της ε, εφημερίας και υπό τη γαλλική νομοθεσία πριν από την απόφαση στην, ε, υπόθεση Γέγκερ, ο χρόνος εφημερίας υπολογιζόταν ως χρόνος εργασίας. Όμως ήταν δυνατό να τον υπολογίσουμε κάτω από 100% ανάλογα με, τον, με, το, με το ποσοστό έντασης της δουλειάς στην περίοδο της εφημερίας. Να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα υπάρχει μια συλλογική ε, συμφωνία ε, που αναφέρει συγκεκριμένο χρόνο εφημερίας, για παράδειγμα 75% του χρόνου εργασίας, για να λάβει υπόψη ε, την τον, την αναλογία ενεργού και ανενεργού χρόνου κατά τη διάρκεια της εφημερίας. Αυτό ε, ήταν γνωστό ως equivalence, ως σύστημα ισοδυναμίας ε, και ειδικότερα σε συλλογικέ συμφωνίες για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ε, σήμαινε νομοθετικό διάταγμα το οποίο ανέφερε συγκεκριμένες διατάξεις συμπεριλαμβανομένων των, συμπεριλαμβανομένων σε βάση της οποίας πρέπει να υπολογίζεται ο χρόνος εφημερίας. Αυτό, επ' Επιλήφθηκε το ε, δικαστήριο στην ε, τελευταία υπόθεση την οποία εκδίκασε. Ε, η απόφαση δημοσιεύθηκε το 2005 αν θυμάμαι καλά. 14 κάθετος 04 είναι ο αριθμός της απόφασης αν δεν απατώμε. Ο υπολογισμός του χρόνου εργασίας δεν θεωρεί συμβατός με, το χρόνο εργασ... με την οδηγία για το χρόνο εργασίας, δηλαδή η αναλογία που χρησιμοποιόταν δεν ήταν η κατάλληλη. Συνεπώς, ο χρόνος εφημερίας θα έπρεπε να θεωρείται 100% χρόνος εργασίας και όχι, το, ως, όχι να υπολογίζεται ως το 75% του χρόνου πραγματικής εργασίας. Δύο σημεία όμως πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με την απόφαση αυτή. Το πρώτο σημείο είναι ότι το δικαστήριο μιλούσε για την εφημερία σε σχέση με το κεκτημένο στο πλαίσιο του, της νομοθεσία. νομοθεσίας και σύμφωνα με τις ε, αποφάσεις ε, ΣΕΜΑΠ και ΓΕΓΕΡ ε, ο χρόνος εφημερίας μπορεί να είναι εκτός του χώρου εργασίας και να υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας υπό την οδηγία. Αν δηλαδή κάποιο είναι σε βάρδια για παράδειγμα στο σπίτι του και πρέπει να πάει να εργαστεί μόνο αν τον καλέσουν τότε αυτό δεν συνιστά χρόνο εργασία. Αυτό το αναφέρει ευθαρσώ η απόφαση ε, ΣΥΜΑΠ ε, Γέγκερ του ε, δικαστηρίου. Όταν όμως δεν παραμένει στο σπίτι ο εργαζόμενος, το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει οι οικογενειακές και επαγγελματικέ ανησυχίες να ληφθούν υπόψη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και συνεπώς σε σχέση με αυτό τον χρόνο εφημερίας, τέλος πάντων συνεχούς βάρδια στο σπίτι, ε, είναι ο χρόνος ε, για τον οποίο καλείται κάποιος να εργαστεί και όντως εργάζεται. Διαφορετικά δεν θεωρείται χρόνος εργασίας. Λοιπόν, ένα σημείο είναι αυτό, ότι ο χρόνος εφημερίας ε, στο χώρο εργασίας είναι 100% χρόνος εργασίας, όμως δεν ισχύει το ίδιο αν η εφημερία γίνεται στο σπίτι, για παράδειγμα. Μιλάμε για το χρόνο εργασίας που περνάει κάποιος στο χώρο εργασίας του. Μόνο αυτός θεωρείται 100% χρόνος εργασίας. Κάτι ακόμη, ο υπολογισμός της, ε, του χρόνου εργασίας το πλαίσιο της οδηγίας για το χρόνο εργασίας, ε, για τον υπολογισμό δηλαδή του ανώτατου ορίου των 48 ωρών, δεν καλύπτει ε, τους, το επίπεδο των μισθών όμως. Συνεπώς, Συχνά οι αναφέροντες ε, διαμαρτύρονται ότι η εφημερία δεν πληρώνεται 100% ε, το ίδιο όσο ο χρόνος πραγματική εργασίας, όμως το δικαστήριο το έχει επιτρέψει αυτό και σε άλλες περιπτώσεις, δηλαδή δεν ισχύει η οδηγία ε, για το χρόνο εργασίας στον μισθό, για το μισθό που καταβάλλεται. αναλύσαμε το νέο διάταγμα του 2009 το οποίο μας γνωστοποίησε ο αναφέρον και, η συλλογική, και τη συλλογική συμφωνία της 4ης Μαΐου 2000 και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι οι εθνικές διατάξεις ακολουθούν ακριβώς ε, αυτό που ζήτησε στην υπόθεση τελάει στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το σύστημα της ισοδυναμίας ε, μπορεί να ισχύσει για τους μισθούς όταν αυτό όμως επιτρέπεται από την κοινοτική νομοθεσία και κατά περίπτωση. Το σύστημα λοιπόν αυτό επιτρέπεται να συνεχίσει να ισχύει για τον υπολογισμό του χρόνου εργασίας μόνο στο βαθμό που αυτό δεν οδηγεί στο να δουλεύουν οι εργαζόμενοι άνω του ορίου των 48 ώρων που θέτει η οδηγία. Η γαλλική νομοθεσία προβλέπει 35 ώρο την εβδομάδα που είναι αρκετά χαμηλότερο από το 48 ώρο που προβλέπει η οδηγία για το χρόνο εργασίας. Το γαλλικό δικαστήριο στην υπόθεση Ντελές ε, εφαρμόζοντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είπε ότι το σύστημα ισοδυναμίας μπορεί να χρησιμοποιείται και στην περίπτωση της ε, ε, εφημερίας στο βαθμό που αυτό ε, που αυτή η εργασία υπερβαίνει το όριο που θέτει ε, η οδηγία για το χρόνο εργασίας. Και είναι σαφές για μας από την εξέταση της νομοθεσίας και της συλλογική ε, συμφωνίας βάσει των στοιχείων που υπέβαλε ο αναφέρον ότι δεν μπορούν να γίνουν περισσότερα για το θέμα αυτό. Για να συνοψίσω, ε, εξετάσαμε πολύ λεπτομερώς όλα τα στοιχεία που ε, μας γνωστοποίησε ο αναφέρον και διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με συμμόρφωση ούτε με την οδηγία ούτε με τις αποφάσεις του δικαστηρίου στις υποθέσεις Γέγκερ και ε, Ντελάς. Το μόνο θέμα που θα θέλαμε να θέσουμε που σε σχέση με την επιχειρηματολογία στην τελευταία επιστολή ε, του αναφέροντος, ο αναφέρον ε, ισχυρίζεται ότι στην πράξη όταν υπολογίζεται ο, ο, ο εβδομαδιαίος μέσος όρος υπηρεσίας των τραυματιοφορέων, δεν εξετάζεται σωστά ε, η το εβδομαδιαίο ρεπό που πρέπει να ε, που προβλέπεται στο πλαίσιο της οδηγίας για τους ε, υπαλλήλους αυτούς. Επίσης υπάρχει και το θέμα των τεσσάρων ε, εβδομάδων ε, άδειας ε, που πρέπει να αφαιρούνται από το συνολικό ποσό όταν γίνεται ο υπολογισμός του μέσου όρου του χρόνου εργασίας. Αυτό είναι αλήθεια, πρέπει να συνυπολογιστεί. Αλλά όπως βλέπουμε από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο, γιατί ο αναφέρον ισχυρίζεται ότι προβλέπεται στον ε, κώδικα ε, εργασίας ε, τη, του γαλλικού κράτους και συνεπώς είναι ζήτημα γαλλικής επιθεώρησης εργασίας. Καλύπτεται από την εθνική νομοθεσία, είναι ένα ζήτημα που αφορά ειδικότερα τον ιδιωτικό τομέα ε, το, τους τραυματιοφορείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και δεν αφορά το θέμα των συλλογικών ε, συμβάσεων ε, γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η συνάδελφος Γκρινή. Ευχαριστώ. Με μεγάλη προσοχή παρακολούθησα και διάβασα αυτήν την αναφορά Και το τελευταίο διάταγμα του 2009 για μένα δείχνει ότι έχουμε πια μπει στο χώρο σεβασμού της οδηγίας για την εργασία, όπως τη γνωρίζουμε. Υπάρχουν οι αντιστοιχίε και για τα άλλα επαγγέλματα, για τους όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Μάλλον δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και πιστεύω θα πρέπει να ισχύει και στο εθνικό δίκαιο και σύμφωνα με την οδηγία. Τα όρια του χρόνου εργασία. 48 ώρες, ναι βεβαίως ένα ζήτημα και ο υπολογισμός της ε, μεταποδοχών άδεια. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι θα πρέπει οι εργαζομένοι, αν διαπιστώσουν ότι στη συγκεκριμένη επιχείρηση για τη νομοθεσία να εντάξει, αν στη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν τηρούνται οι ε, διατάξει νομοθεσία, θα πρέπει να αντιδράσουν. Και ναι, μπορεί να λέει η επιχείρηση, α, δεν προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε, αλλά αν έρθει ένα εργαζόμενο να καταγγείλει ε, παραβάση της νομοθεσίας, ε, παραβίαση νομοθεσίας σχέση με το χρόνο εργασίας, τότε συνήθως αναλαμβάνει τη σχετική δράση. Για μένα πρέπει να κλείσει η αναφορά. Έχει δοθεί η απάντηση. Φυσικά δεν είμαστε θέση να γνωρίσουμε αν αυτά που μας ε, επισημαίνουν οι αναφερόμενοι ευσταθούν ή όχι, αλλά για τη Γαλλία πιστεύω ότι η Γαλλία θα πρέπει να ρυθμίσει τα θέματα αυτά εσωτερικά πλέον. Για τις αμοιβές είχε και το ίδιο. Ότι οδηγία δεν προβλέπει τίποτα για αμοιβέ. Και ως εκ τούτου, εδώ αναγκαστικά παραπέμπουμε στις, στις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς στη Γαλλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Ποστινάρο θέλει να παρέμβει, όχι. Ο αναφέρον θέλει κάτι να προσθέσει. No. Non c'è una replica da parte Φαίνεται πως όχι. Άρα παραμένει ανοιχτή η αναφορά. Με συγχωρείτε, κλείνουμε, κλείνουμε την αναφορά όπως ε, ζητήθηκε. Περνάμε στο, στην αναφορά υπαριθμών 12 που υποβλήθηκε από έναν πολίτη ισπανικής ηθαγένειας σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών στη Ναβάρα, δυνάμει της Οδηγίας 2003-88 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν το λόγο έχει η κυρία από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορούμε πιο σύντομη σε σχέση με αυτή την αναφορά. Δεν έχουμε νέα στοιχεία. Είχαμε δώσει μια ανακοίνωση το 2008, τον Νοέμβριο. Δεν μας έχει ενημερώσει με άλλο τρόπο ο αναφερόμενος. Και η θέση μας είναι αυτή την οποία είχαμε εκφράσει και το 2008, τα κύρια στοιχεία δηλαδή που αναφέρει αναφερόμενος, είναι πως η εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης μπορεί να μεταφερθεί στην προσεχή εβδομάδα. Στην Αβάρα για τους αστυνομικούς ισχύει αυτό. Αυτό ρητά το προβλέπει η οδηγία και προβλέπει και εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης, όμως το άρθρο 68 λέει ότι αυτή η εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης μπορεί να μετακυληθεί στην επόμενη εβδομάδα. Και με τη νέα οδηγία μπορεί τους ή άλλου να μετακυληθεί ακόμη περισσότερο, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας. Σας ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, ε, παρεμβάσεις αντιρρήσεις ως προς το κλείσιμο. Φαίνεται ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να αποφασίσουμε υπέρ του κλεισίματος αυτής της αναφοράς. Περνάμε στην επόμενη, υπάρχει 13, είναι παρόν ο αναφέρον ή όχι. Η κυρία Σαντάλ Πόνς, εξ του αναφέροντος. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι ο αναφέρον ε, λυπάται ιδιαίτερα διότι δεν του δόθηκαν τα στοιχεία, δεν του διαβιβάστηκαν τα στοιχεία από το γαλλικό κράτος. Ε, με βάση τις 18, τα στοιχεία της 18 Φεβρουαρίου 2010. Και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για στελέχη που έχουν ε, δυνατότητα λήψη αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 17 της οδηγίας. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα εξή Η γαλλική αστυνομία είναι ένα ιεραρχικό σώμα με βάση τρία ε, σώματα. Το σώμα πλαισίωσης και εφαρμογής που αφορά ενωματάρχες και αξιωματικούς, το ε, δεύτερο σώμα που εκπροσωπεί 11.500 και το σώμα, το διευθυντικό σώμα το οποίο περιλαμβάνει τους ε, γενικούς επιθεωρητές που εκπροσωπούν 1.800 υπαλλήλους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε να κάνουμε με μία ενδιάμεση διαβάθμιση. Δεύτερον, υπάρχουν, ε, υπάρχει μία διαδικασία που αναφέρεται στα αντίστοιχα, ε, στα αντίστοιχα σήματα ανάλογα με το κάθε σώμα. Τρίτον, ο ορισμός των αποστολών καταδεικνύει ότι υπάρχει μία ιεραρχία διότι η δυνάμη του άρθρου 2 της, του διατάγματος 2005-716 σε σχέση με το, την πρώτη διαβάθμιση του σώματος αυτού δείχνει ότι αναφέρεται στο ότι θα μπορεί κανείς να υποκαταστήσει τους ε, επιθεωρητές. Τέταρτον, αυτό τονίζεται ακόμα ακόμα περισσότερο από την αποστολή των επιθεωρητών αστυνομίας που θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας και καλύπτουν οργανικές θέσεις. Πρόκειται για το άρθρο 2 του Διατάγματος 2005-939 της ε, Δευτέρας Αυγούστου 2005 σε σχέση με το, σώμα, το Διευθυντικό Σώμα της Εθνικής Αστυνομίας. Το 6% των αξιωματικών αστυνομίας διέπονται από το άρθρο 4 του Διατάγματος 2815 σε σχέση με τη μείωση χρόνου εργασίας στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή ε, σε σχέση με την εβδομαδιαία εργασία και δεν έχουν καμία ε, αυτονόμηση διαχείρισης. Το υπόλοιπο 4 διέπεται από το άρθρο 10 του εν λόγω διατάγματος σε σχέση με τη διαχείριση χρόνου εργασίας με βάση την πλαισίωση των επιθεωρητών αστυνομίας. Ας λάβουμε υπόψη την απόφαση του ΔΕΚ, υπόθεση σε 484 κάθετος 04, Επιτροπή κατά Ηνωμένου Βασιλείου. Εξαίρεση δυνάμει του άρθρου 17. Άρα πιστεύω ότι οι διάφορες διαβαθμίσεις ε, επιθεωρητέων και μη ε, εντάσσονται σε ένα ιεραρχικό πλαίσιο δυνάμει της, ε, και εντάσσεται στη διεύθυνση των επιθεωρητών αστυνομίας. Άρα διέπονται από το άρθρο 17 ένα στοιχείο α της οδηγίας, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τους αξιωματικούς υπηρεσίας. Ζητάμε λοιπόν ε, η, ώστε η γαλλική νομοθεσία να διέπεται από την οδηγία 2003 κάθετος 88 κάθετος ΕΚ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να παρέμβουν οι συνάδελφοι. Οι εκπρόσωπες της Επιτροπής σας έχω το, δώσει το λόγο τόσες φορές που είχα την εντύπωση ότι σας τον έδωσα και τώρα ζητώ συγγνώμη. Δεν υπάρχει πρόβλημα κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ναι, πολύ ευχαριστώ να δώσουμε την ενημέρωση και ταυτόχρονα στήσουμε συγγνώμη στον αφαιρόμενο που δεν έλαβε λεπτομερή ενημέρωση από την ε, πλευρά μας για την αναφορά του. Πρόκειται εδώ για την εφαρμογή της οδηγίας για το χρόνο εργασία στη Γαλλία σε επίπεδο κατώτερων στελεχών της ε, Εθνικής Αστυνομίας Πολύ Νασιονάλ. Εδώ έχει γίνει σχετική αλλαγή για τον χρόνο εργασία. Κάποια από τα προβλήματα που επισημαίνουν οι αναφερόμενοι, ποσοστά αμοιβών για τι υπερορίε ή για απασχόληση έξω από το πεδίο τη οδηγία. είναι έξω από το πεδίο τη οδηγία, ναι, όπως εξήγησα και νωρίτερα, αλλά έχουμε επίση την απάντησή μα, του Ιανουαρίου 2010 πώ εξακολουθούμε να έχουμε να τρέφουμε ανησυχίες ως σε, σε σημεία που επισημαίνει ο Διότι υπάρχουν κάποια ζητήματα ευθυγράμμιση στην οδηγία, καταρχάς όσον αφορά το ουσιαστικό όριο για την ετήσια περίοδο απασχόληση. για το λεγόμενο αυτό corps de τους υπαξιωματικούς, και δεύτερον, ε, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, εάν δεν υπάρχει αποτελεσματικό όριο εργασίας την εβδομάδα, ξεπερνάμε το χρόνο εργασίας που επιτρέπεται ανά εβδομάδα από την οδηγία. Η οδηγία με το άρθρο 17.1 προβλέπει τη δυνατότητα παρέκκλησης για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίοι μπορούν αυτόνομα να ε, ορίσουν το χρόνο απασχόλησης τους. Το επίπεδο τώρα, το ιεραρχικό αυτού του κόρτου κομμανού στη γαλλική αστυνομία δεν ξέρουμε αν υπάγεται πράγματι στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Έχουμε αμφιβολίε για το κατά πόσο υπάγεται. Έχουμε αναπτύξει άτυπες μέχρι στιγμής ε, συνομιλίες με τι εθνικέ αρχέ, οι οποίε μέχρι στιγμή δεν έχουν διασκεδάσει τι αμφιβολίε που είχαμε εκφράσει στι ε, παρατηρήσει μα. Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε μια λεπτομερή απάντηση και πάλι όταν λάβουμε την επίσημη απάντηση από τις γαλλικές αρχές. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορούσα να δώσω πιο πολλές πληροφορίες. Επιβεβαιώνω όμως ότι διατηρούμε τις αμφιβολίες που είχαμε εκφράσει στην προηγούμενη μας απάντηση. Και περιμένουμε από τις εθνικές αρχές. Ο κύριος Κυρία Πρόεδρε, κοιτάξτε, εδώ είναι σαφές. Η αναφορά πρέπει να παραμείνει εκρεμής μέχρι να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τις αρμόδιες αρχές της Γαλλίας για το πώς έχουν τα πράγματα. Οπότε προτείνω να παραμείνει ανοιχτή η εν λόγω αναφορά. Ε, η κυρία Γκρουνή. Συμφωνώ απολύτω γιατί νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφεί οι απαντήσει. Είναι περίπλοκο γιατί εντάξει, εγώ δεν γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς ε, είναι οι βαθμίδες των αστυνομικών. Ε, γνωρίζω το δίκαιο της εργασίας ε, στον ιδιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, για το διευθυντικό στέλεχος μιας επιχείρησης. Υπάρχουν διάφορες βαθμίδες και υπάρχουν μάλιστα και ορισμένες θέσεις εργασίας που είναι αρκετά αυτόνομες. Οπότε όταν χρειάζεται κάποιο να δουλέψει περισσότερο, υπάρχει αντιστάθμιση με κάποιο χρόνο ανάπαυση. Εγώ διάβασα τα έγγραφα και δεν είναι σαφέ, είναι γεγονό ότι δεν είναι σαφέ ε, σε σχέση με την αποζημίωση. Αν υπάρχουν δηλαδή κατά αποκοπήν ποσά ε, προς συγκεκριμένες ε, βαθμίδες του αστυνομικού ε, σώματος ανάλογα με το χρόνο εργασίας τους. Ίσως λοιπόν πρέπει να μείνουμε ανάλογα, να, μείνουμε, να μείνει ανοιχτή η συγκεκριμένη αναφορά μέχρι να έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει να απαντήσει ο εκπρόσωπος του αναφέροντος για ένα λεπτό. Ναι, κοιτάξτε, δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω, πολύ απλές. Ε, στην επιστολή του 2008 του Διευθυντή της ε, Αστυνομίας είναι ότι δεν ε, υπάρχει κανένα ωράριο για τους αστυνομικούς, δηλαδή αυτή τη στιγμή όμως στο πλαίσιο της οδηγίας ε, είναι απολύτω πιθανό να γνωρίζει κανείς ακριβώς πόσες ώρες ε, δουλεύει. Δεύτερον, έχει γίνει αναθεώρηση και συνεπώς είναι πάρα πολύ εύκολο να γνωρίζουμε κατά πόσο ένας αστυνομικός ε, ή κάποιος ανώτερος του έχει κάποια διευθυντική εξουσία, κάποια εξουσία απόφασης ή όχι. Είναι πάρα πολύ σαφές τι συμβαίνει και είναι δύο παρατηρήσεις που θα ήθελα η Επιτροπή σας να λάβει υπόψη. Και εμείς θα αποτανθούμε στην Εκτελεστική Επιτροπή διότι θα πρέπει να μπει στη διαδικασία επαλήθευσης και γι' αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία ε, του αναφέροντος. Άρα η αναφορά παραμένει ανοιχτή και θα δούμε τι θα γίνει με τις επόμενες φάσεις. Η τελευταία είναι του Ζων Πιρότ και του δίνω το λόγο. Je Σας ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς το γαλλικό κράτος ε, είναι ε, σε κατάσταση παράβασης διότι δεν εφαρμόζει τον, τον κανονισμό και το διάταγμα της 14ης Δεκεμβρίου 2000 έχει ψηφιστεί εδώ και 9 χρόνια, όμως δεν έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, ιδιαίτερα όσον αφορά το άρθρο 24. Από το 2006, επειδή δείξαμε μεγάλο ενδιαφέρον για τις οδηγίες και την ε, εφαρμογή τους, Μάθαμε για την ύπαρξη του κοινοτικού δικαίου και είδαμε ότι ε, πολλοί πυροσβέστες δεν εντάσσονταν σε αυτό το πλαίσιο. Και γι' αυτό θα πρέπει να, μας, να αναλάβουμε υπόψη ότι πολλά δημοτικά συμβούλια έχουν μεταφέρει την οδηγία αλλά δεν την εφαρμόζουν και δυστυχώς ε, επιτελείται μαύρη εργασία με τη συγκατάβαση των ε, εθνικών αρχών. Δυστυχώς όμως οι πυροσβέστες πρέπει να τύχουν προστασία σε δύναμη των οδηγιών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η οδηγία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άρα θα πρέπει να δούμε τους επαγγελματίες και μη που θεωρούνται ε, εθελοντές. Δεν είναι εθελοντές, διότι ο Βελικός νόμος της 3ης Εβδόμου 2005 ορίζει τον εθελοντισμό ως δραστηριότητα η οποία δεν αμείβεται. Ο αριθμός των επαγγελματίων αφορά μια σύμβαση πενταετή η οποία είναι ανανεώσιμη και ο μη επαγγελματικό τομέα αφορά μια σύμβαση, μια πενταετή σύμβαση η οποία είναι ανανεώσιμη. Πρόκειται για ένα 99% δραστηριότητας ε, όπου υπάρχουν ίδιες αποστολές, ε, οι ίδιες, ε, τα ίδια ωράρια, διατρέχουν τους ίδιους κινδύνους και αν λάβουμε υπόψη το βασιλικό διάταγμα της 3ης Ιουνίου 1999 βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με την ίδια εργασία. Δεν πρέπει να ε, ξεχνάμε, και τις ειδικέ δραστηριότητες ως προς το χρόνο εργασίας. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το διάταγμα Γέγκερ της 9ης ε, 2003 που ε, ενέκνε και το ΔΕΚ. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για την παρουσία τους στις συγκεκριμένες ε, ζώνες κινδύνου. Άρα, οι μη επαγγελματίες πυροσβέστες δεν έχουν κανένα περιορισμό στο χρόνο εργασίας και θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες εβδομαδιαίως, 168 ώρες εβδομαδιαίως χωρίς διακοπή ο επαγγελματικός κλάδος που τηρεί την ε, οδηγία και τις 38 ε, ε, νόμιμες ώρες δεν την χάνει της ίδιας μεταχείρισης, διότι ένας εργοδότης μπορεί να επιβάλλει το ίδιο πλαίσιο για τους επαγγελματίες και μη, τη στιγμή που μιλάμε για σόρευση 168 ώρων. Άρα οι μη επαγγελματίε την χάνουν διάκριση διότι εντάσσονται στην ίδια υπηρεσία και διατρέχουν τους ίδιους ε, κινδύνους ατυχήματο. Το ίδιο αφορά και το συνταξιοδοτικό, γιατί στην περίπτωση των μη επαγγελματιών δεν εντάσσονται στο ε, εθνικό πλαίσιο συνταξιοδότησης. Με βάση την εφαρμογή της οδηγίας κάθε κάθετος 104, επειδή δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, κάθε μέρα διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο ως πυροσβέστες και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει παραβίαση του κοινοτικού δικαίου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την προσοχή σας. Υπάρχουν παραβιάσεις της τάξης των 15 με 16.000 ημερησίως. Ευχαριστώ πολύ και δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Thank you, Madam President. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι η μόνη από τις ε, αναφορές που έχουμε σήμερα όπου δεν έχουμε δώσει γραπτή ανακοίνωση. Γιατί θα πρέπει, προκειμένου να το πράξουμε αυτό, να διευκρινίσουμε ορισμένα από τα περιστατικά αυτής της υπόθεσης από αυτά που βλέπουμε σήμερα στην αναφορά είναι πολύ δύσκολο να κρίνουμε σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο και σε ποιο βαθμό δεν εφαρμόζεται. Να σας εξηγήσω γιατί. Ο ανεφερόμενος λέει ότι οι εθελοντές πυροσβέστες, πυροσβέστες δηλαδή προσλαμβάνονται με διαφορετικούς όρους από τους επαγγελματίες έχουν, ε, είναι στη διάθεση, υπηρεσία του 168 ώρες την εβδομάδα. Αυτό είναι το συνολικό ε, διάστημα διαθεσιμότητας, εφημερίας, αν θέλετε, την εβδομάδα ε, σε ημέρες και σε σύνολο ημερό, και σε σύνολο εβδομάδας. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο διάστημα παραμένουν στην υπηρεσία κατά την οποία θα έπρεπε όλο αυτό το διάστημα να υπολογιστεί ως χρόνος εργασίας με βάση και την οδηγία ή αν πρόκειται απλώς για χρόνο στον οποίο, κατά τον οποίο βρίσκονται στο σπίτι τους αλλά σε επιφυλακή και στη διάθεση υπηρεσίας, εάν τυχόν προκύψει κάποιο κατεπηγόν περιστατικό. Εάν συμβαίνει αυτό η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη με βάση και ε, τη σχετική απόφαση του δικαστηρίου. Διότι τότε μόνο όταν κληθούν ε, στην ε, δουλειά τους θα υπολογιστεί αυτός ο χρόνος, ως χρόνος απασχόλησης, χρόνος εργασίας. Άρα πρέπει να ξέρουμε αν έχει χρόνος κατά τον οποίο είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στον χώρο εργασίας, αν έχουν φερειπίν υποχρεωτική κατάρτιση κατά τη διάρκεια των ορών αυτών, εάν η περίοδος αναφοράς είναι μία εβδομάδα, και αν κάθε εβδομάδα υπάρχει αυτός ο χρόνος απασχόλησης, αν είναι ο μέσος όρος απασχόλησης ανά εβδομάδα, αν είναι ο μέσος όρος απασχόλησης σε περίοδο ενός έτους και ούτω καθεξής. Είναι πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να ε, διευκρινιστούν. Μας λέει ο αναφερόμενος ότι απασχολούνται και άλλου. Ναι, πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν πόσες ώρες απασχολούνται στην άλλη τους εργασία. Για δε ορισμένα από τα θέματα τα οποία προκύπτουν ε, στην αναφορά μπορεί να βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας όπως είδαμε και σε προηγούμενες απαντήσεις, φερειπίν ζητήματα των τιμολογίων για την αποζημίωση ή της διαφοράς ε, μεταχείρισεως μεταξύ των επαγγελματιών πυροσβεστών και των εθελοντών. Ή τα θέματα της ασφάλισης, ε, κάλυψης των ε, εργασιακών ατυχημάτων κτλ. Ξέρουμε ότι πρόκειται για ένα τομέα κρίσιμο για την δημόσια ασφάλεια. Έχουν να κάνουν με πολύ δύσκολες καταστάσεις οι πυροσβέστες και πρέπει να εξασφαλίζεται η κατάλληλη περίοδος ανάπαυσης. Τόσο για το δικό τους καλό, όσο και για το καλό των πολιτών που περιμένουν τη βοήθειά τους σε μια περίπτωση ανάγκης. Θα θέλαμε όμως να διευκρινιστούν όλα αυτά τα σημεία πριν να δώσουμε μια πιο οριστική απάντηση στην υπόθεση αυτή. Υπάρχουν πολλά ασαφή σημεία ε, κεντρική σημασία στην την άποψή μα ε, και εκεί δεν μπορούμε να δώσουμε επαρκή ε, απάντηση. Στο συγγνώμη, λυπούμε. Αν είχαμε πιο πολλέ γραπτέ πληροφορίε για τα σημεία αυτά, θα μπορούσαμε να λύσουμε την κατάσταση και να δώσουμε μια λεπτομερή απάντηση. Φαντάζομαι θα ήταν πιο χρήσιμη. Ο κύριος Μποστινάρη. Με καταπλήσετε Μπορεί να φταίει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο κοινοβούλιο και τη βελγική κυβέρνηση και δεν έχει φτάσει μέχρι εδώ η απάντησή τους. Αν και ήξερα ότι λειτουργεί το ταχυδρομείο στο Βέλγιο. Δεν ξέρω πώς τελικά παραπέμπονται στις καλένδες οριστικά αυτές οι απαντήσεις από τη βελγική κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει όμως έχουμε να κάνουμε ένα συγκεκριμένο πρόεδρο, ε, πρόβλημα. Πρόεδρε πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό και έχει υποχρέωση η εθνική κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά από τη δική μου πατρίδα, από τη ρουμανική κυβέρνηση και τη στάση τη κυβέρνηση τη Ρουμανία, ότι ακολουθεί ακριβώ την ίδια μεθοδολογία. Αλλά παραμένει πρόβλημα. Πρέπει να του πείσουμε με κάποιο τρόπο να δίνουν απαντήσει σε ερωτήσει μα. Διότι χωρί απάντηση τη βελγική κυβέρνηση, πώ μπορούμε είτε να διαπιστώσουμε παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων και ως εκ τούτου να αναλάβουμε πέρα το δράση ή να διαπιστώσουμε ότι είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία οι βελικοί κανόνε, εφαρμόζονται ορθά από τη βελική κυβέρνηση και ω εκ τούτου σταυρώνουμε τα χέρια και δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά είναι τώρα πολύ ασαφή η κατάσταση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να αποστείλουμε μια θερμή επιστολή στη βελγική κυβέρνηση και ίσως να βρούμε κάποιον ε, υφυπουργό που να βρίσκεται ακόμη εν ζωή και να είναι σε θέση να μας δώσει απαντήσει. Ο αναφέρον θέλει κάτι να προσθέσει. Μπορεί ίσως και εκείνος να μας αποστείλει ένα γραπτό υπόμνημα, αν θέλει, στη συνέχεια. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ πολύ σύντομα να πω ότι οι εθελοντές περασβέστες ε, εργάζονται 102 ώρες εφημερία την εβδομάδα και το μήνα με τέσσερις ε, ομάδες που εναλλάσσονται στις βάρδιες τους 168 ώρες όπως είπαμε είναι παρόντες ανα πάσα στιγμή είναι στη διάθεση της υπηρεσίας σε μία ζώνη δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ε, παραμονή κατοίκων πρέπει να βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή που ορίζεται σε μια ζώνη, είτε είναι στο σπίτι τη θιά του, τη γιαγιά του, πρέπει να είναι μέσα σε πέντε λεπτά στην έφεση τη υπηρεσία. Είναι μια συγκεκριμένη ζώνη. Και μάλιστα οι περισσότερε κοινότητε ε, για να σας αποδείξω ποια είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, δεν έχουν σχετικό ε, οίκημα ε, μέσα στο οποίο να στεγάζονται οι πυροσβάσεις, κατά την περίοδο της ε, εφημερίας αυτής. Άρα βρισκόμαστε μέσα σε μια ζώνη διαθεσιμότητας προς την υπηρεσία. Είναι υποχρεωμένες οι κοινότητες να ε, κρατήσουν σε μια ε, ζώνη, όπως είπα, δεσμευμένους για να μπορούν να μας καλέσουν όποτε χρειάζεται. Δεν μπορούμε ούτε σινεμά να πάμε, δεν μπορούμε ούτε με τα παιδιά μας να ασχοληθούμε, ούτε στο σπίτι μας να γυρίζουμε να μακριά και το καθεξής. Ο εργοδότης επίσης είναι ο ίδιος πρέπει να πω με, τους επαγγελμα... Ε, με, την άλλη εργασία. Δηλαδή είναι η δημόσια υπηρεσία ε, του Δήμου, καλύτερη υπηρεσία του Δήμου, η οποία του ε, βάζει να δουλεύουν το πρωί και το βράδυ είναι σε εφημερία ω εθελοντέ πυροσβέστε. κοιμήθηκαν δεν κοιμήθηκαν. Αν την άλλη μέρα το πρωί που θέλουν να ξαναπάνε στο γραφείο για την άλλη του δουλειά ε, είναι ξενυχτισμένοι γιατί χρειάστηκε να κάνουν παρέμβαση σε μια περίπτωση πυρκαγιά, ε, τότε κάκο του κεφαλιού του. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι η κυβέρνηση του Βελγίου μα έχει ε, αντιμετωπίσει με γη αλλά εάν θέλει βεβαίως πιο λεπτομερή ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πολύ ευχαρίστω. Δεν ήμουν σίγουρα ότι θέλατε τόσο